την εισηγήτρια τη Επιτροπή Προπολογισμών, την κυρία Αντρέασεν τη Επιτροπή Προπολογισμών, για να δούμε κατά πόσο οι διαπιστώσει τη θεμελιώνονται. Διότι η εικόνα που έχουμε εμεί για τον τομέα τη Αλία είναι τελείω διαφορετική από εκείνη που περιγράφει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα γενικευμένο πολιτικό πρόβλημα επί του πέραν των όσων θα συζητήσουμε σήμερα. Τώρα επί της ουσίας. Ζήτησα σήμερα να βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνεδρίου και γι' αυτό ζήτησα τον κύριο Λαζάρου να είναι μαζί μας. Γιατί έχω την αίσθηση, όταν διάβασα δηλαδή την έκθεση και τη μελέτησα προσεκτικά, και μπορέσαμε να αντιθούμε ατύπω και με εκπροσώπου του Ελληνικού Συνεδρίου. Είχα τέλο πάντων την αίσθηση ότι η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου από τη μια εισάγει στοιχεία απολύτω ορθά τα οποία έχουν να κάνουν με τη λογιστική λειτουργία του ίδιου του συνεδρίου. Από την άλλη όμως εισάγονται και στοιχεία αποτίμηση που θα έπρεπε να είναι τη αρμοδιότητα ενό νομοθέτη. το ελληνικτικό συνέδριο δεν είχε καμία διάθεση να παρέμβει σε αρμοδιότητε νομοθετικέ, βεβαίω. Αλλά περισσότερο αφοσιώσαμε την προσοχή μα στο να δούμε πώ αυτή η έκθεση που εντοπίζει την ανεπάρκεια των μέτρων για τη διάλυση έχει πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. μάλλον στόχος δεν ήταν ε, η ε, κατάρρευση, αλλά ακριβώς η μείωση των ελεκτικών ικανοτήτων. Το Ελεκτικό συνέδριο μας λέει ότι το αποτέλεσμα δεν έχει επιτευχθεί. Και συμπεραίνει ότι δεν το διαθέτουμε, δεν το έχουμε, δεν έχουμε μελλοντική στρατηγική που να μπορέσει να προβλέψει μελλοντικές παρεμβάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για την διάλυση σκαφών. Στο σχέδιο έκθεσης που έχετε μπροστά σας, όπου χρειάστηκε βεβαίως και θα χρειαστεί να επιφέρω κάποιες αλλαγές μετροπολογίες που θα υποβληθούν, και ανάλογα και με τις συζητήσεις, τις διαρκείς συζητήσεις όπως εξελίσσονται και τις συνομιλίες μας από το ελεκτικό συνέδριο. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή έχει και κάποια όρια. Τα όρια αυτά είναι κατά πρώτον ότι αξιολογεί τη γενική κατάσταση. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά βάσει της εντολής που έλαβα. Η αξιολόγηση λοιπόν είναι γενική και αφορά το σύνολο, τη συνολική εικόνα των ευρωπαϊκών δράσεων. Δεν υπάρχει επαρκής διάκριση ανάλογα με τις περιοχές ή τις κατηγορίες αλίας. Υπάρχει λοιπόν μια ομογενοποίηση ενώ σε μερικές περιοχές της ευρωπαϊκή Ένωσης η διάλυση ήταν ε, ε, αποτελεσματική απάντηση για, την, ε, για τον περιορισμό των στόλων, σε άλλες περιοχές αυτό δεν συνέβη. Το να καταλήγουμε λοιπόν σε ένα απλό συμπέρασμα και να γίνεται αυτό αποδεκτό, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ταυτόχρονα την ιδέα, την ιδέα τη ε, τυπική προσέγγιση ότι αυτό είναι ένα δρόμο που δεν μπορούμε πλέον να προκρίνουμε. Κάτι που δεν ταιριάζει και με την ε, νομοθετικού και πολιτικού περιεχομένου συζήτηση που μπορεί να γίνει σε μια επιτροπή όπω η δική μα. Αυτό, όπω είπα, είναι μια προσέγγιση λογιστική. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρξει αποτίμηση πολιτική. Διότι το αποτέλεσμα στην Ευρώπη είναι διαφορετικό από μέρο σε μέρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η διάλυση δεν λειτουργούσε πουθενά. Όχι. Άλλε περιοχέ ε, ανέτρεξαν στην διάλυση, άλλε όχι άλλες λιγότερο, άλλε περισσότερο. Αυτές είναι οι, γενικές ε, παρατηρήσεις, η πρώτη γενική παρατηρήση που είχα να κάνω. Η δεύτερη παρουσιάζει και αυτή ένα πρόβλημα. Η έκθεση αναφέρει για το μέλλον ότι οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνονται στην μεταβιβασιμότητα των αδειών, των δικαιωμάτων. Και αυτό γίνεται με τοποθέτηση, κατά τη δική μου άποψη, πάλι πολιτική. Δηλαδή, ε, λογιστική εξέταση του όλου θέματος. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καταδεικνύουμε αυτή την προσπάθεια ως μόνη οδό για την μείωση των, ε, της των αλληλευτικών στόλων. Δεν είναι μόνο η μεταβασιμότητα των δικαιωμάτων, διότι επανελειμμένο ζήτησα από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας προσφέρει αποδεκτικά στοιχεία ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να συνεισφέρει στο μέλλον στην μείωση των αλληλευτικών προσπαθειών. Κανεί από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να μου το αποδείξει τελικώ. Αυτέ σε γενικέ γραμμέ λοιπόν είναι οι δικέ μου θέσει ω προ την έκθεση. Ήταν ε, προσοδοφόρα η συνεργασία μας με το ελεγκτικό συνέδριο. Συναντηθήκαμε και ατύπως και επισήμω και οι απόψεις μας όσο και αν μεταβλήθηκαν ελαφρώς, οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Υπήρξε ασάφεια της εντολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ελληνικό Συνέδριο. Γι' αυτό τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης κάποιες φορές δεν ε, μας βρίσκουν σύμφωνους. Γι' αυτό λοιπόν με κάποιες τροπολογίες σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να μετατραπεί, να μεταβληθεί η εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ελληνικό Συνέδριο. Ίσως έτσι να καταφέρουμε να διευκρινίσουμε καλύτερα το αποτέλεσμα που θα προσδοκούμε. Τα πρώτα εδάφια της εκθεσής μου, που είναι σύντομη αλλά ελπίζω περιεκτική, θα λάβουν υπόψη το είδος εντολής που θα λάβει το ελεγκτικό συνέδριο διότι πιστεύω ότι μεταξύ άλλων στην έκθεση αναφέρονται και διαφορετικές λύσεις. Όχι με σαφήνεια βέβαια, αλλά η δράση του ελεγκτικού συνεδρίου επικεντρώθηκε σε ένα μόνο στοιχείο. Το κατά πόσον θα είναι τα μέτρα αυτά αποτελεσματικά. Όμως, στο κείμενο της έκθεσης μεταξύ άλλων αναφέρονται και κάποιες επιπλέον λύσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη. Αυτή λοιπόν η δική μου ημέρημνα προκύπτει από το γεγονός, και αυτό το έχω διευκρινίσει, ότι όποια και είναι η κατάληξη των δικών μας συζητήσεων, δεν θα πρέπει να προκαταλάβουμε τις εργασίες μας για τη μεταρρύθμιση διότι έτσι θα αντιφάσκαμε με την ε, εντολή μας. Το λέω αυτό σεβόμενος ε, καθόλου τις ε, τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχει και η Λισαβόνα η οποία ανέθεσε στους βουλευτές το κοινοβούλιο μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Όποιο λοιπόν και αν είναι το συμπέρασμα, όποια και αν είναι η κατάληξη της συζήτησης για την νομοδότηση και ελπίζω να διορθωθεί έτσι και η γενική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου που λέει κάποια πράγματα παράλογα για τον τομέα μας. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ένα μήνυμα που θα επηρεάσει τις εργασίες που γίνονται είτε για τον βασικό κανονισμό είτε για την ουσία του Ταμείου αλλά ούτε και για το υπόλοιπο των εργασιών μας. Είναι μια κρίσιμη έκθεση. Ο χαρακτήρας της είναι κρίσιμος. Και βεβαίω εδώ ουσιαστικά εμπεριέχεται και το πνεύμα μια προσωπικότητα του Κοινοβουλίου που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μιλάνα. Κύριε Λαζάρο, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Κύριε Μιλάνα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. και ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλάνα που βρήκατε χρόνο για μας. Έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά βρήκατε χρόνο να συζητήσετε την πρότασή σας για σχέδιο γνωμοδότησης σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Αρχίζοντας, θα ήθελα να πω ότι το έργο του ελεκτικού συνεδρίου είναι να ελέγχει την, το πώς εκτελείται ο προϋπολογισμός και να φέρει στην προσοχή των νομοθετικών αρχών οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν. Στην περίπτωση αυτή, διεξάγαμε ελέγχου στα υπάρχοντα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χωρητικότητα των αλληλευτικών στόλων και τις αλληλευτικές ευκαιρίε. Λάβουμε την εντολή από την ε, συνθήκη και έτσι λοιπόν ούτε η Επιτροπή ούτε κανένας άλλος δεν μας έδωσε εντολή να διεξάγουμε αυτή την έρευνα. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας έκθεσής μας για τα μελλοντικά ε, έργα που θα αναλάβουμε, συμπεράναμε ότι αυτή η περιοχή μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία στους ε, ενδιαφερόμενους αλλά και για τις νομοθετικές αρχές. Ιδιαίτερα μάλιστα διότι η κοινή αλληλευτική πολιτική γινόταν, θα έφτανε σε σημείο αναθεώρησης. Το ελεκτικό συνέδριο ως εκ τούτου δεν κάνει συστάσεις για πολιτική. Και όχι μόνο σε αυτήν εδώ την ειδική έκθεση, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη ειδική έκθεση. Οι συστάσεις πολιτικής δεν είναι τμήμα της εντολής μας και πέραν αυτού όταν ένας εξωτερικός ε, ελεκτής κάνει συστάσεις πολιτικής σημαίνει ότι είναι μέλος της ε, εκτελεστικής εξουσίας, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και μάλιστα τόσο πολύ ώστε εάν αυτές οι πολιτικές δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα τότε ο εξωτερικός ελεκτής, στην περίπτωση αυτή τον, το ελεκτικό συνέδριο, είναι μέρος της διαδικασίας αυτής. Δεν είναι αυτό όμως το έργο μας. Το έργο μας είναι να δώσουμε σε εσά την το νομοθετικό όργανο, τα εργαλεία για να συζητήσετε και να λάβετε τις πολιτικές αποφάσεις που είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε θέμα, με οποιοδήποτε θέμα ασχολείστε αυτή τη στιγμή, εν προκειμένου την κοινή αλληλευτική πολιτική. Και το πρόβλημα της ε, βιώσιμης αλληλείας. Κατόπιν τούτου, θα ήθελα να σχολιάσω τις συστάσεις μας όσον αφορά τις μεταβιβα... τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Δεν δεν πρεσβεύουμε ότι αυτά τα δικαιώματα είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα. Απλά θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι η Κομισιόν πρέπει να αποσαφηνίσει ότι οι άδειε αυτές μπορούν να μειώσουν, ε, να, ελαττώσουν το πρόβλημα. Και αυτό το αναφέραμε, διότι ο ισχύων κανονισμός δίνει αντιφατικά μηνύματα για τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα και αναφέρομαι στην παράγραφο 28 της ειδικής μας έκθεσης όπου τονίζουμε ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ε, σε περίπτωση που τα αλληλευτικά δικαιώματα πρέπει να αποσύρονται κτλ. κτλ. Αυτός ο κανονισμός για ε, απόσυρση αντέρχεται σε άλλο σημείο του κανονισμού. Επίσης, ο λόγος τον, για τον οποίο αναφερθήκαμε στα μεταβάσιμα αλληλευτικά δικαιώματα είναι ο εξής. Σε μία από τους χώρους που επισκεφτήκαμε, την Δανία, στο, στα επιχειρησιακά τους ε, προγράμματα είχαν συμπεριλάβει τα, τις ε, μεταβιβάσιμες αλληλευτικές άδειες. Και σύμφωνα με τις δανεικές αρχές, κατάφεραν να μειώσουν τον αλληλευτικό στόλο κατά 27% ανάμεσα στο 2003 και το 2009, χωρίς δημοσίες δαπάνες, χρησιμοποιώντας απλά αυτές τις μεταβιβάσιμες άδειες. Στην παράγραφο όμως 33 τονίζουμε ότι η πρακτική αυτή στη συγκεκριμένη χώρα και σε μία άλλη, την οποία επισκεφθήκαμε, είχε να κάνει με ειδικέ περιπτώσεις αλίας που δεν είναι ίδιες με τις μικτές ε, περιπτώσεις που υπάρχουν σε άλλα ευρωπαϊκά ύδατα και αυτές οι, αλλα... Ε, οι επιλογές ήταν επιλογές των συγκεκριμένων κρατών μελών για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό το αναφέραμε και επαστήσαμε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους και κάναμε σύσταση στην Κομισιόν να διασαφίσει εάν αυτό είναι κάτι που, μπορεί, μπορούν, να που μπορούν να κάνουν και στη συνέχεια, αν θα μπορούσε να είναι μια λύση στο πρόβλημα. Όσον αφορά το σχέδιο για τα σκάφη για τη διάλυση σκαφών. Πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο δεν κατάφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρότι καταβλήθηκαν προσπάθειες. Συμφωνώ πόλητα με τον κύριο Μιλάνα ότι ο έλεγχος ασχολήθηκε με το συνολικό πρόβλημα και δεν επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες μορφές αλίας. Από την άλλη όμως κατά τη διάρκεια των ελέγχων μας, εάν είχαν προκύψει ζητήματα σχετικά με την σημασία συγκεκριμένων τύπων αλίας, αυτά τα έχουμε αναφέρει στην έκθεση. Είμαι στη διάθεσή σας τώρα για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Και στα αριστερά μου έχω τον κύριο Κοντρία, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας ε, που διεξήγαγε τον έλεγχο. Εγώ λοιπόν και ο κύριος Κοντρία είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Λαζάρου. Θα έχουμε ένα γύρο ερωτήσεων τώρα με τους ευρωβουλευτές, ο κύριος Στίβεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μιλάνε και κύριε Λαζάρου για τις παρουσιάσεις αυτές. Δέκα περίπου χρόνια πριν Όταν χρησιμοποιούσαμε τις επιχορηγήσεις για την ναυπήγηση νέων σκαφών, αποφασίστηκε από την πλειοψηφία αυτής εδώ της Επιτροπής ότι η πρόταση του να χρησιμοποιηθούν λεφτά των φορολογούμενων για να διαλυθούν ορισμένες φορές καινούργια αλλιευτικά σκάφη και ε, να διαλυθούν γιατί οι διοκτήτες τους δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνεια για αυτά τα σκάφη. Και τα μεγάλα σκάφη έχετε υπόψη ότι κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ και διαλύονταν αυτά τα σκάφη με χρήματα των φορολογούμενων σε, ένα, σε ορισμένα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χρήματα των φορολογούμενων είχαν χρησιμοποιηθεί για να ναυπηγηθούν καινούργια σκάφη. Καταλήξαμε ότι αυτή η πρακτική δεν ήταν καθόλου βιώσιμη και κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών να καθυστερήσουν όλες οι σχετικές επιχορηγήσεις και να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον μόνο για ορισμένες πτυχές ε, εξυγχρονισμού για να βελτιωθεί ασφάλεια στα σκάφη. Και αυτή ήταν η σύσταση της Επιτροπής και του ΕΤΑ για την ε, μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Ξέρω ότι ο κύριος Καντέκ θα ήθελε πολύ να επανεισαγάγει τις επιχορηγήσεις για την ε, ναυπήγηση και, την, και τον εξυγχρονισμό των σκαφών και αυτό πιστεύω ότι θα μας πήγαινε προς τα πίσω. Όμως, πριν από λίγες εβδομάδες ήμουν στην Βόρεια Ιρλανδία σε ένα από τα μικρότερα λιμάνια με στόλο περίπου 30 ετών σε ηλικία και μου είπαν λοιπόν ότι ναι, εάν δεν μας αφήσετε, εάν δεν μας επιχορηγήσετε να σε νέων σκαφών τουλάχιστον πρέπει να μας επιτρέψετε να έχουμε αλλιευτικές παραχωρήσεις για τα επόμενα χρόνια. Γιατί τότε θα μπορούμε να πάμε με αυτό στην τράπεζα και να δανειστούμε το 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ που χρειαζόμαστε για να αναφυγήσουμε ένα νέο αλλιευτικό σκάφος. Και αυτό το επιχείρημα είναι πολύ σωστό. Είναι βασικό. Και αυτό πιστεύω ότι προτείνει και η Κομισιόν στο νέο πακέτο μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Εάν λοιπόν επιτρέψουμε στους αλληλείς, στους ίδιους τους αλληλείς να επενδύσουν στην αυπήγηση νέων αλληλευτικών σκαφών, χρειαζόμαστε αυτές τις παραχωρήσεις ή με περιορισμούς μεταφοράς ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μπορούμε να τους κάνουμε θελοντικούς, ε, τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά και πριν. Δεν μπορούμε όμως να κρατάμε δύο καρπούς για κατά από την ίδια μας χάλη σε αυτή την περίπτωση ή να κάνουμε αυτό με το οποίο διαφωνώ έντονα, να επιχορηγήσουμε τις ναυπηγήσεις νέων σκαφών που νομίζω κιόλας ότι δεν θα αντιμετωπίσει την ε, πλεονάζουσα αλληλευτική δυνατότητα ή να ε, εισαγάγουμε τις παραχωρήσεις με ειδικού όρους. Ευχαριστούμε κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου γιατί πραγματικά μας ε, την προσοχή στις αδυναμίες του ε, σχεδίου. Παρόλες τι αδυναμίες όμως, το σχέδιο αυτό λειτουργεί και δυστυχώς ενδεχομένω να αυξήσει την ε, αλληλευτική ικανότητα παρά να τη μειώσει όπως είναι επιθυμητό. Πιστεύω ότι το ε, επεξηγηματικό σημείωμα ε, λαμβάνει μια έντονη θέση και την υπερασπίζεται έντονα, πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Μιλάνα είπε κάτι πολύ σωστό για τις διαφορές ανάμεσα στους τύπους αλίας και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το σύστημα και διαφορετικές συνθήκες σε κάθε κρατός μέλος. είχα όμως, έχω όμως δύο ερωτήσει. στους ελεκτές και ίσως τον κύριο Μιλάνα. Πρώτο το θέμα της πλεονάζουσας ε, λευτικής ικανότητας. Συζητήσαμε χθε σε αυτή την επιτροπή και υπόθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ότι δεν έχουμε αυτή την πλεονάσια ικανότητα. Ο δικός σας ορισμός από πού προκύπτει. Ή ενδεχομένω. ή να έχετε λάθος από την αρχή δηλαδή λέγοντας ότι υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα στον ευρωπαϊκό στόλο. Άρα λοιπόν έχετε αρχίσει λάθος στην έκθεση. Να το δούμε αυτό. Έπειτα, αυτό που είπε ο κύριος ε, Μιλάνα, ότι ζητά να χορηγηθούν κονδύλια με δύο τρόπους. Και για να ε, υποστηρίξουν μέτρα για τα πληρώματα που υφίστανται συνέπειες ε, στην, με τη διάλυση των σκαφών. Φυσικά, συμπονώ με αυτούς τους ελείς. Οι καπετάνοι όμως ε, έχουν κερδίσει, κερδίζουν αρκετά χρήματα. Τα πληρώματά τους όμως είναι αυτά που υποφέρουν. Δεν έχω καταλάβει όμως γιατί θα έπρεπε να χορηγηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια με αυτά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κλείνουν μαγαζιά αυτή τη στιγμή για, για χαμηλή ζήτηση, ε, λόγω της ύφεση και πολλά καταστήματα επίσης ε, γίνονται διαδικτυακά. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί δεν επιχορηγεί, δεν αποζημιώνει τους καταστηματάρχες. Καταλαβαίνω πολιτικά ε, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της αλληλευτικής πολιτικής πώς ε, λειτουργεί αυτό, αλλά δεν είμαι και τόσο... Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δώσει ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτή την αλλαγή. Μου φαίνεται κάπως μου φαίνεται ότι δεν σέβεται τους ε, κανόνες των επιχειρήσεων. Και μετά θεωρεί το ελεκτικό συνέδριο, οι ίδιοι ελεκτές, ότι αυτή είναι σωστή χρήση των κονδυλίων για βιομηχανική αλλαγή στα, στα αλληλευτικά σκάφη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Μιλάνε για την έκθεση και χαίρομαι και για την ε, έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που εστιάζεται στα στρεβλωτικά μερικές φορές ε, αποτελέσματα που είχε το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Ταμείο στην προηγούμενη περίοδο. Και μία φράση τα λέει όλα. Από την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2002 τα ελιεύματα έχουν μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο τόνους και έχουν χαθεί ε, περίπου 100.000 θέσει απασχόλησης. Νομίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα υπερβολικής γενεοδορίας και επιδαψίλευσης κονδυλίων για να παραμείνουν πολλοί στην αλία και να ψαρεύουν ένα όλο και πιο περιορισμένο αριθμό αλληλευτικών αποθεμάτων. Το θέμα είναι Ποιο είναι ο ορισμό της πλεονάζουσας ελευτικής ικανότητας. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε την πλεονάζουσα ελευτική ικανότητα. Όταν δεν μπορεί καν να βγάλει το ψωμί του από, το, από την αλίευση ο ψαράς, πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει πλεονάζουσα ελευτική ικανότητα. Φαίνεται ότι ο ελευτικό κλάδος δεν συμβάλλει στο αέρα. Τα κέρδη του αλληλευτικού κλάδου είναι πολύ χαμηλότερα από τα κονδύλια που χρειάζονται για να στηριχθεί αυτός ο κλάδος. Δεν είναι και πολύ θετικά αυτά τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια ικανότητας, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου τη γνώμη του γι' αυτό γιατί το ελεκτικό συνέδριο ανισχύει τα ανώτατα όρια ελευτικού στόλου προκειμένου να μειωθεί ε, ο ελευτικός στόλος είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο, μια και ε, το μέγεθος του ελευτικού στόλου και το ανώτατο όριο είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος του ίδιου του ελευτικού στόλου, οπότε δεν έχει περιοριστικό αποτέλεσμα το ανώτατο όριο στις διαστάσεις τελικά στο μέγεθος του ελευτικού στόλου. Οπότε το Ελεκτικό Συνέδριο πρότεινε τι μεταβάσεις με σε ελευτικές άδειες ως τρόπο, για μείωση, του ελευτικού στόλου. Αλλά πώ θα ελέγξουμε πραγματικά την ελευτική ικανότητα σε κάθε κράτο. και πιστεύω ότι θα μπορεί να, θα μπορεί να μειωθεί ο ελευτικός στόλος με τη μείωση του ανώτου του όριου ε, ελευτικής ικανότητα. και αν ναι, γιατί δεν ήταν πιο αυστηρή η σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου αν θεωρεί το μέτρο αποτελεσματικό, γιατί ουσιαστικά το άφησε στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών το θέμα της μείωσης του αλληλευτικού στόλου. Συμφωνώ με τον κύριο Στίβενσον ότι θα πρέπει να είναι προαιρετικό αυτό το σύστημα για τα κράτη-μέλη, αν θέλουν να εισαγάγουν αυτές τις ε, μεταβιβάσιμες ελευτικέ άδειες θα πρέπει να είναι κούσιο το σύστημα και να υπάρχει και ένα όριο ε, κοινοτικό σε ό,τι αφορά την ε, ικανότητα, την αλληλευτική ικανότητα. Ο κύριος Γκάλαχερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και τον κύριο Μιλάνα για τα σχόλιά τους. Συμφωνώ καταρχήν με τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι το μητρό στόλο, το νεολόγιο, θα πρέπει να ενημερώνεται σωστά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η βάση. Αν δεν έχουμε λεπτομέρειες του Μητρώου του Νεολογίου σε κάθε κράτος, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πλεονάζωσης ικανότητας. Το Μητρό είναι η βάση για τον έλεγχο. Και όταν πρωτοθεσπίσαμε τα Μητρώα, μερικές χώρες ήταν πολύ πιο έξυπνες και δεν έκαναν και πολλά. Και η ελευτική τους ικανότητα ήταν πολύ χαμηλότερη. Ενώ χώρες που ήταν πιο έντυπες, και έδιναν τα σαφή στοιχεία για τον αριθμό του, των ελευτικών σκαφών βρέθηκαν χαμένες τελικά. Δεν ήταν επαρκής ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μητρό, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Γι' αυτό και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, επειδή ακριβώ υπήρξαν ανεπάρκειες τότε. Θα πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση του Μητρό Ελευτικών Σκαφών σε ό,τι αφορά την πλεονάζουσα ικανότητα. Τι θα πει πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα. Είναι πολύ φλού αυτό το θέμα, πολύ γενικό και όριστο. Δώστε μου ένα παράδειγμα να το καταλάβω. Αν πάρουμε τα πελαγικά σκάφη, θεωρούμε ότι τα σκάφη ε, αλλιεύουν 365 μέρες το χρόνο. Τώρα, ό,τι και να ψαρεύουν, σκουμπρί, ρέγγα, Σαρδελόρεγκα, ο αριθμός είναι περιορισμένος. Στα πελαγικά σκάφη, έξι μήνες το χρόνο, ψαρεύουν πολύ λιγότερο. Θεωρητικά όμως, κατά 50% παρουσιάζουν πλεονάζουσα ηλεκτρική ικανότητα. Παρόλο που για το δεύτερο εξάμεινο δεν υπάρχουν ε, πελαγικά είδη να ψαρέψουν. Στα χαρτιά υπάρχει πλεονάζουσα λευτική ικανότητα, αλλά αυτά τα σκάφη τα χρειαζόμαστε για να ψαρέψουν έστω και το μισό χρόνο. Γιατί το προσφυγάκι, τη ρέγκα, ε, το σκουμπρί δεν τα βρίσκουν ε, τα λευτικά σκάφη όλο το χρόνο, παρά μόνο το μισό. Προσοχή λοιπόν τι επιχείρημα χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό της πλεονάζουσας ελευτικής ικανότητας. Και επίσης, προσοχή κύριε Μιλάνα. Μία από τις συστάσεις σας λέει, θεωρεί ότι οι μεταβιβάσιμες ελευθερικές άδειες είναι η μοναδική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος πλεονάσεως ικανότητας. Δεν είναι η μοναδική λύση, κύριε Μιλάνα. Μπορεί να αποτελεί τμήμα της λύσης, αλλά σίγουρα δεν είναι η μοναδική λύση. Α, συγγνώμη, το ελεκτικό συνέδριο το λέει Σύντο συγγνώμη από τον κύριο Μιλάνα. Το ανακαλώ. Την τελευταία φορά που είχαμε ακρόαση με τον ε, εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου ήταν πολύ ρεαλιστική, αντικειμενική, αλλά με ανησυχεί αυτό το σχόλιο του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι οι μεταβιβάσιμε ε, ελευθερικέ άδειε είναι η μοναδική λύση για τον έλεγχο τη πλεονάζουσα ικανότητα. Δεν συμφωνώ με αυτό δεν πιστεύω ότι είναι τεκμηριωμένο και φαίνεται ότι δεν υπάρχει σωστή αντίληψη του προβλήματος. Και ε, όταν Μάρθα Μάντερσον μας ε, συμβουλεύει για τα ευρωπαϊκά θέματα, ε, είμαστε επιφυλακτικοί γιατί γνωρίζουμε τις θέσεις της. Πάντως, επαναλαμβάνω, το μητρό ελευτικό σκαφό θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και σωστά. Συμφωνώ με τον Στρουέν Στίβενσον. Το βασικό ζήτημα είναι η ασφάλεια. Αν έχουμε σκάφη 25-30 χρονών και μερικά είναι και ακόμη πιο παλιά, δεν μπορούν να, να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τους αλείς να επαναφέρουν τα σκάφη τους στις προδιαγραφές ασφάλειας. Επίσης, αν έχουμε ένα πλοίο κατάστρωμα, θα πρέπει να γίνει πιο ασφαλές. Πώς θα το καταστήσουμε ασφαλές, θα κλείσουμε κάπως το κατάστρωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιορίζουμε την ε, ικανότητα του αλληλευτικού σκάφους, απλώς το κάνουμε πιο ασφαλές. Δεν νομίζω ότι έτσι περιορίζουμε ή αυξάνουμε με τις προδιαγραφές ασφάλειας την ικανότητα ή την αλληλευτική δυνατότητα πλεονάζουσα ικανότητα διαφέρει το σε άλλος από χώρα σε χώρα και από, από αλληλευτικό είδος σε αλληλευτικό είδος. Δεν ξέρω, καλό ή κακό υπάρχουν τέτοιε διαφορέ. Θέλουμε λοιπόν διευκρινήσει για αυτά τα σημεία. Κύριος Φεραίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να βλέπουμε την αλία ως κάτι παραπάνω από ένα απλό εμπορικό τομέα. Ένα χώρο συναλλαγών όπως οποιοδήποτε άλλος. Διότι εδώ υπόκειται και ένα άλλο θέμα μεταξύ όλων αυτών που συζητούμε. Γιατί τελικώς αποζητούμε να έχουμε μια κοινή και πολιτική. Εάν πιστεύουμε ότι αυτή η αλληλευτική πολιτική πρέπει να επιδιώκει στόχους όπως ε, το κοινό συμφέρον, όπως η κάλυψη των επιστημιστικών αναγκών του πληθυσμού, η ανάπτυξη της απασχόλησης, η προστασία των ε, παράκτιων κοινοτήτων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε γιατί να επιδιώκουμε και να πετύχουμε τους στόχους αυτούς θα πρέπει η πολιτική να πρικοδοτηθεί με τα απαραίτητα μέσα ακόμα και σε δημοσιονομικό επίπεδο η αγορά θα διαδραματίσει εδώ έναν ρόλο σε όλα αυτά. Καταλήγουμε να συζητούμε όλους αυτούς τους στόχους ε, σαν κάτι που να διέπεται μόνο από την αγορά. Ενώ από δημοσιονομικής άποψης ε, και από κάθε άλλη δεν πρέπει να βλέπουμε απλώς την αλία σαν έναν επιπλέον εμπορικό τομέα. Ως προς τους χαρακτηρισμούς για το στόλο. Το πρόβλημα είναι ότι κάποια πράγματα γίνονται παραδεκτά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα πράγματα για το χαρακτηρισμό του στόλου. Δεν μπορούμε να παραμένουμε σε γενικόλογους και επιφανειακούς χαρακτηρισμούς για την πλεονάζουσα ικανότητα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι στόλοι υπάρχουν, ποιοι έχουν την πλεονάζουσα ικανότητα, για ποια είδη, σε ποιες περιοχές, σε ποιες γεωγραφικές ζώνες. Αυτές τις απαντήσεις αναζητούμε και σήμερα δεν είμαστε σε θέση να τις δώσουμε. Το αναγνωρίζει και η ίδια Επιτροπή. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να βρούμε απαντήσεις σε ένα προσεχές μέλλον. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά. Ε, και επιμένω, δεν μπορούμε να μετατρέψουμε την πραγματικότητα που σε μεγάλο βαθμό είναι παραγνωρισμένη δεν μπορούμε να την αγνοούμε σε βαθμό που να μην συνάδει με τους στόχους που επιδιώκουμε. Θα ήθελα ο συνάδελφος Μιλάνα στην έκθεση του να εισαγάγει κάποιες προτάσεις σημαντικές θεωρώ. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αποζημίωση για τους ε, που χάνουν τη ε, δουλειά τους λόγω διάλυσης σκαφών. Δεν υπάρχουν προγράμματα κοινωνικής προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για όποιον ε, χάνει τη δουλειά του. Αυτό εντάξει είναι κάτι που ισχύει, αλλά δεν είναι λόγος αυτός για να το εισάγουμε και στον χώρο της αλίας, επειδή υπάρχει σε άλλους τομείς. Στην περίπτωση της αλίας θα έπρεπε εδώ να υπάρχει κοινοτικοποίηση κάποιων ε, συστημάτων. Αυτό θα πει κοινή πολιτική αλίας, ε, να υπάρχει και κοινό πολιτικό κόστος. Γιατί θέλουμε κοινή πολιτική αλίας μόνον για να υπάρχει η ελευθερία στα κάτι μέλη να αναπτύσσουν όπως θέλουν την κοινή ελευθερική τους πολιτική και το κόστος πρέπει να το μοιραζόμαστε. Δεν μπορεί να είναι μόνο εθνικό. Εάν υπάρχει κοινή πολιτική θα πρέπει να μεταφράζεται ακριβώς και στην πράξη και στο τομέα του κόστους. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστο αυτή τη κοινή ελεκτική πολιτική, δηλαδή να αποζημιώνονται όσοι χάνουν τη δουλειά του λόγω διάλυση σκαφών. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω είναι σημαντικό να εμφανιστεί στην έκθεση Μιλάνα. Και κάτι άλλο, μια άλλη σημαντική παρατήρηση που κάνατε κι εσεί. και θα τη συναντήσουμε και αργότερα. Η διάκριση που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μεταξύ αλληλευτική ικανότητα και αλληλευτική προσπάθεια, δυνατότητα Εδώ το γεγονό ότι υπάρχει μείωση τη αλληλευτικής ικανότητα δεν σημαίνει ότι υπάρχει και μείωση τη αλληλευτικής δυνατότητα, της προσπάθειας. Εδώ, αν σκεφτούμε τι γίνεται με τι μεταβεβαίσιμε άδειε ε, στι αζόρε, θα δούμε ότι είναι κάτι που πολλέ φορέ δημιουργεί προβλήματα. Η μείωση τη αλληλευτικής ικανότητα, εφόσον ε, εφαρμοστεί το σύστημα των μεταβεβάσιμων αδειών, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα υπάρξει και ε, περιορισμό τη αλληλευτικής προσπάθειας θέλουμε να μην σκεφτόμαστε τα πράγματα μόνο από οικονομική πλευρά και μόνο από τον οικονομικό ανταγωνισμό. Κάποιοι θα καταστραφούν και αυτοί που θα μείνουν τελικά θα ψαρεύουν όσο και προηγούμενοι και όσο όλοι μαζί. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και συγκέντρωση τη αλληλευτική προσπάθεια χωρί να υπάρχει τελικά μείωση τη αλληλευτική ε, ε, το αποτελέσματο. Εδώ και το ελεγκτικό συνέδριο το λέει αυτό για το σύστημα μεταβιβάσιμων αδειών. Ε, ότι είναι μια επιλογή πολιτική, μια πεποίθηση. Και θα τεθούν πολλά προβλήματα με την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Δεν έχουμε ακόμη εμπειρία από αυτή την πρακτική. Δεν ξέρουμε στην πράξη τι θα γίνει, οπότε τίποτε δεν μας εγγυάται ότι το σύστημα αυτό είναι λύση και μάλιστα πανάκια ίσα ίσα που μπορεί και να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φεραίρια. Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Ε, thank you, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε εδώ να περιοριστούμε στο να πούμε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στην Επιτροπή σας, ότι καλωσορίζουμε τα συμπεράσματα της ειδική έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Και απλώς να πω ότι η συμφωνία αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνο σε όλα τα σημεία. Συγκεκριμένα, η πλεονάζουσα ικανότητα καταμετράται καθημερινά από τα κράτη-μέλη. Όμως, η ποιότητα των εκθέσεων των κρατομελών δεν είναι ακόμη ικανοποιητική. Βελτιώνεται, αλλά δεν είναι ακόμη αρκετή. Ούτε επαρκής. Αυτή είναι η εξήγηση για το ότι δεν έχουμε μια σαφή απάντηση για το τι γίνεται με την της ικανότητα ανά ε, στόλο και ανά περιοχή αλίευσης. Ευχαριστώ κύριο Λαζάρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Ελίας για τις ερωτήσεις τους. Τη σημείωσα. Και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Αν στην πορεία χρειαστώ κάποιες διευκρινήσεις για ορισμένες ερωτήσεις, θα σας ε, υποβάλω συμπληρωματικές ερωτήσεις. Καταρχήν να δώσω μια απάντηση στα σχόλια του κυρίου Φερέιρα και του κύριου Γκάλεχερ. Το ελεκτικό συνέδριο είπατε ότι πιστεύει πως η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι η θέσπιση του συστήματος μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων ή αδειών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν υποβάλλει τέτοια σύσταση. Δεν ε, είναι αρμοδιότητα του ελεκτικού συνεδρίου η υποβολή συστάσεων του ελεκτικου συνεδριου υποβολη συστασεων πολιτικης Απλώ προέκυψε στη διάρκεια του ελέγχου και επιστήσαμε την προσοχή των ενδιαφερομένων και των νομοθετικών αρχών σε αυτό το θέμα. Και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα μεταβιβάσιμων αναλυτικών αδειών θα διαδραματίσει ποιο ρόλο. Αλλά δεν ε, τασόμαστε εμεί υπέρ τη θέσπιση ενό τέτοιου συστήματο, το θεωρούμε μοναδική λύση. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει του κυρίου Ντέιβι η πρώτη ερώτηση για την πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα και το κατά πόσο υπάρχει καταρχήν τέτοια. Η απάντηση, η απάντησή μου είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη του μεγέθους της πλεονάζουσας ικανότητας. Και όπως αναφέρεται στην παράγραφο 73 της έκθεσης, ε, εξαιτία πλημελού ενημέρωση ε, και χορήγηση στοιχείων από τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει σαφή αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ισορροπία μεταξύ αλληλευτικής ικανότητας και αλληλευτικών δυνατοτήτων. Κάτι που ε, δυσκολεύει την εφαρμογή πολιτικών για την μείωση της πλεονάσεως ικανότητας και την αξιολόγηση των επιδόσεων τέτοιων πολιτικών. Τούτο λεχθέντος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο της έκθεσης που επισημαίνει ότι την τελευταία φορά που αποτιμήθηκε η πλεονάζουσα ικανότητα ήταν ε, το 95, και όταν δόθηκε το ποσοστό το 40% της πλεονάσματος. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Τα ελιεύματα από 7 εκατομμύρια το 1995 μειώθηκαν σε 5 εκατομμύρια το 2009. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ελευτικού στόλου, υπήρξε μια μείωση από 100.000 πλοία το 1995 σε 1,8 εκατομμύρια τόνους ή 80.000 ελευτικά σκάφη το 2009. Από 2 εκατομμύρια τόνους σε 1,8 από 100.000 σκάφη σε 80.000. Αλλά χρειαζόμαστε ακριβείς πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για να αποτιμήσουμε το επίπεδο πλεονάζωσης ικανότητας. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα, ως προς τη δεύτερη ερώτηση του κυρίου Ντέιβις. Αν δεν κάνω λάθος, αφορούσε την επιχορήγηση για την ε, ανασυγκρότηση, τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, μπορείτε να την επαναλάβετε. Ναι. Το θέμα είναι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ΕΤΘΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, για να αποζημιώσουμε πληρώματα σκαφών που πάβουν την αλληλευτική του δραστηριότητα υπόκειται σε διάλυση και άρα οι ναυτικοί μένουν άνεργοι. Είναι αλήθεια ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι μια κοινοτική, ενωσιακή πολιτική και άρα φέρουμε ιδιαίτερες ευθύνες ε, για την αλληλεία σε σχέση με άλλους ε, οικονομικούς ε, κλάδους. Και φαντάζομαι ότι οι πλειοκτήτες θα αποζημιωθούν. Αν μη τι άλλο με την επιδότηση της διάλυσης ή από αν δεν μπορέσουν να απολύσουν τις ποσοστώσεις τους. Αλλά τα μέλη του πληρώματος θα χάσουν τη δουλειά τους και το μέλλον του θα είναι ζωφερό. Θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια του ΕΤΘΑ για την αποζημίωση των πληρωμάτων. Αλλά δεν μπορούμε ε, ταυτόχρονα να αποζημιώνουμε και άλλου ε, εργάτες ε, οποιοδήποτε βιομηχανικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που μένουν άνεργοι. Γι' αυτό διαρωτώ με ένα σκόπιμο να χρησιμοποιούμε κοινωτικά κονδύλια για τέτοιου είδου αποζημιώσεις. Ένα προβληματισμό έθεσα στον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν είμαι υπέρμαχο τη μία ή τη άλλη λύση ο κύριος Λαζάρο. Ευχαριστώ κύριε Ντέβις. Η απάντησή μου δυστυχώς είναι ότι δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δεν είναι αρμοδιότητα του ελεκτικού συνεδρίου η χάραξη πολιτικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χρήματα των φορολογουμένων και το κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για παροπλισμό, διάλυση πλοίων ή για τον εξυγχρονισμό ε, των πλοίων ή επενδύσεις ε, για επενδύσεις στα πλοία, τι να σας πω. Δεν πρόκειται το ελεκτικό συνέδριο να επικρίνει πολιτικές επιλογές. Εμείς απλώς σχολιάζουμε την αποτελεσματικότητα τέτοιων επιλογών. Για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι ε, η χρήση του συστήματος ε, της διάλυσης θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένο. Γιατί φαίνεται ότι δόθηκαν κονδύλια για παροπλισμό πλοίων που ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Ίσως δεν πληρούνται τα κριτήρια ε, για τον παροπλισμό συγκεκριμένων πλοίων, άρα θα κακώς δόθηκαν κονδύλια. Τώρα, για τις επενδύσεις ε, στα πλοία, πάλι με κρατικά, με κοινοτικά κονδύλια. Είπαμε ότι επειδή οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την αλληλευτική ικανότητα των πλοίων, θα πρέπει να επαναξεταστεί αυτό το σύστημα, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της αλληλευτικής ικανότητας του πλοίου με τη χρήση τέτοιων κρατικών κονδύλιων κοινοτικών. Καλώς. Ο κύριος Μιλάνα τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Νομίζω η συζήτηση αυτή συνεισέφερε στο να διευκρινιστούν ένα-δυο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, από το ελεγκτικό συνέδριο δεν έρχεται καμία ένδειξη που να μας λέει ότι το σύστημα μεταβιβάσιμων αδειών είναι λύση. Ίσα ίσα στο άρθρο 30 της έκθεσης, πολύ σαφώς λέγεται και το παραθέτω, για να υπάρξει μείωση της αλληλευτικής ικανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα, πολιτικά μέσα. Αυτό αποδεικνύει το σύστημα των μεταβιβάσιμων αδειών αλληλεύσης μπορεί να είναι μια αποτελεσματική απάντηση για την τη αλληλευτικής ικανότητας, αλλά δεν είναι η μόνη και δεν είναι μια απόλυτη αλήθεια. Αυτό το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο. Επίσης καταγράφουμε το γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι δεν είναι δυνατό να ορίσουμε την πλεονάζουσα ικανότητα. Δεν υπάρχουν εργαλεία, δεν υπάρχουν μέσα που να μας, ε, επιστημονικά, τα οποία να μας επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Εάν ε, θέλετε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι επαρκτό γεγονό η πλεονάζουσα ικανότητα. Όμω αυτό μπορεί να το δει κανεί με λεπτομέρειε στι διάφορε γεωγραφικέ περιοχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με κατηγορία αλληλεία. Μόνο στην πράξη. Και το συζητήσαμε και χθε. Τα όρια που αναφέρει το ελληνικό συνέδριο στο άρθρο 73 της έκθεσης και σε σχέση με την έλλειψη δεδομένων, αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν να ακολουθήσουμε την προτροπή του κυρίου Καντέκ, το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την ε, συλλογή δεδομένων, να φτάσει στο 75%. Είναι, μια μάχη που έχει δει ο κύριος Φερέρα σε άλλες περιπτώσεις, αλλά το θεωρώ αναγκαίο για να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς. Και κάποιες ε, παρατηρήσεις για την όλη συζήτηση επί της ουσίας. Υπάρχει εδώ ε, η δυνατότητα να είναι αποτελεσματική η διάλυση και να είναι συνεπείς οι πολιτικές μας επιλογές και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της αλίας. Δεν μιλάμε για μια γενικευμένη διάλυση, αλλά ένα πρόγραμμα στοχευμένο σε συγκεκριμένε διαλύσεις. Δηλαδή να μην ε, δαιμονοποιηθεί η διάλυση, αλλά εάν υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ συγκεκριμένο, πολύ ειδικό και εκεί μπορούμε να καταμετρήσουμε και τον αντίκτυπο. Εκεί μπορούμε να σχεδιάσουμε και συγκεκριμένα προγράμματα, στοχευμένα. Στην βασική έκθεση του Ταμείου για την Θάλασσα και την Αλία, δεν θα προβλεφθεί αυτό βέβαια, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στοχευμένα προγράμματα για τη διάλυση μπορούν να, ε, να οργανωθούν και μπορούν και να υλοποιηθούν. Τώρα, για τη φιλοσοφική συζήτηση, το αν θα πρέπει να αποζημιώνονται οι άλλοι, δηλαδή να έχουμε και μια κοινωνική μέρημνα για τους εργαζομένους, νομίζω επ' αυτού θα πρέπει, θα πρέπει να υπάρξει μια υγιής realpolitik από δικής μας πλευράς. Κύριε Λαζάρου, Δίκαιο έχετε ότι δεν μπορεί να απαντήσει στο θέμα αυτό το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι πολιτικού χαρακτήρα το θέμα. Εγώ όμω από πολιτική άποψη ρωτώ το Κοινοβούλιο. Πότε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τη απόφασής μας θα επηρεάσουν όχι την αγορά, καλά λέει ο κύριος Ντέιβις, αν επρόκειτο για την αγορά, θα ήταν η αγορά εκείνη που θα έπρεπε να υποστεί τι συνέπειε ή μια χώρα από την ε, απόλία τη απασχόληση. Αλλά ποια είναι η δική μας επιλογή, γιατί αυτά είναι η υλοποίηση της, δικής, της πολιτικής που σχεδιάζουμε, είναι η ευρωπαϊκή πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι μια χωρα απο την απωλεια της απασχολησης αλλα ποια ειναι η δικη μας επιλογη γιατι αυτα ειναι η υλοποιηση της δικης της πολιτικης που σχεδιαζουμε ειναι ευρωπαικη πολιτικη νομιζω λοιπον οτι μια σκεψη μια εικόνα φιλελεύθερη για όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο, στο νου μας. Διότι με τις διαλύσεις σκαφών προφανώς εντωμεταξύ οι πλειοκτήτες βρήκαν απόκριση στην μειωμένη κερδοφορία τους. Και τελικά βρεθήκαμε με αλληλείς οι οποίοι δούλευαν στα σκάφη, οι οποίοι μάλλον δεν ε, σταμάτησαν να δουλεύουν, απλώς υπήρξε κοινωνικός αντίκτυπος. Δηλαδή από το ένα σκάφος πέρασαν σε άλλα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να συλλογιστούμε να μην τα βλέπουμε τα πράγματα μαύρα ή άσπρα. Να σκεφτούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της επιλογής μας, όχι του γενικότερου σχεδιασμού. Διότι εδώ δεν καθορίζουμε την πολιτική της αυτοκινητοβιομηχανίας που μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο νοσοκροστασίου και να βρεθούν ε, απολυμμένοι τόσοι εργαζόμενοι. Όχι, αυτά τα χρόνια ε, ε, προβλέψαμε δράσεις πολύ στοχευμένες, συγκεκριμένες. Τα λέγαμε, διάλυσε το σκάφος, άσε τις απευθύνσουν σε άλλα αποθέματα, όμως ξεχάσαμε ότι τα σκάφη αυτά δεν τα δούλευαν μόνο ο πλειοκτήτης, αλλά και οι εργαζομένοι του. Ο πλειοκτήτης λοιπόν καλύφθηκε, δεν καλύφθηκαν όμως οι εργαζόμενοι, οι αλληλείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτοί στην προσέγγιση μας, να ακούμε όλες τις απόψεις. Δεν είναι δημοκρατική προσέγγιση εδώ. Πρέπει απλώς να σκεφτόμαστε ότι κάποια αποτελέσματα προκύπτουν από δικές μας πολιτικές επιλογές. Και κλείνω με μια τελευταία παρατήρηση. Ολοκλήρωσα, ολοκλήρωσα. Ε, μια ερώτηση για τον Πρόεδρο. Αύριο λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Νομίζω ότι το καλύτερο ήταν να πάμε ως την Τρίτη την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας ή δυνατόν. Διότι το πρωί δεν συζητήσαμε ακόμη την έκθεση της ε, ε, Επιτροπής Προπολογισμών. Εγώ θα συναντήσω την εισηγήτρια της Επιτροπής Προπολογισμών την Τρίτη. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Ήξερα ότι ο κύριο Ντέβι θα υποβάλει ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πρόβλημα. Να προτείνουμε η διορία να παραταθεί μέχρι την Τετάρτη, 12 το μεσημέρι. Εντάξει. Παράταση προθεσμίας μέχρι την Τετάρτη, Τετάρτη ή 4 Ιουνίου. momento. Bien, me dicen que no es posible adelantar. Μου, μου λένε ότι το πολύ μέχρι τη Δευτέρα επιτρέπεται παράταση. Μέχρι τις 4 Ιουνίου δηλαδή, όχι την Τετάρτη. Αλλιώς δεν προλαβαίνουμε να μεταφράσουμε. Δεν θα προλάβουμε να μεταφράσουμε τις τροπολογίε. Parece que puede haber problemas para traducir. Μάλλον θα υπάρξουν προβλήματα με τη μετάφραση. Οπότε παρατείνουμε μέχρι τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου. Μέχρι τις 4 Ιουνίου παρατείνεται η διορία για την υποβολή τροπολογιών. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης, όπως είχαμε συμφωνήσει. Στο σημείο 9 δηλαδή, την έκθεση Φερέρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαζάρο που ήρθε να μας παρουσιάσει τη γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σημείο 9 για την ερασιτεχνική παραδοσιακή ελεία και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο δεν είχαμε προλάβει, δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Το Μάρτιο είχαμε παρουσίαση της έκθεσης και τον Απρίλιο του σχεδίου της έκθεσης. 7 Μαΐου έληξε η προθεσμία για τις τροπολογίες. Κατατέθηκαν 214 τροπολογίες για το σχέδιο έκθεσης. Η Επιτροπή Ρέγγι ε, Περιφερειακής Πολιτικής και η Επιτροπή Γυναικών επίσης υπέβαλαν τις γνωμοδοτήσεις τους. Τώρα έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας για μια γενική επισκόπηση των τροπολογιών και τι διαπραγματευτικές δυνατότητες έχουμε για να μέσα σε συμβαστικέ τροπολογίε ω προ το σχέδιο έκθεση. Το λόγο έχει ο συγγητή ο κ. Φεραίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τις πολυάριθμες τροπολογίες. Ε, αρκετές από αυτές, όλες μάλλον, δείχνουν το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτή την έκθεση. Ο αριθμός τους το αποδεικνύει αυτό. Και επιβεβαιώθηκε η απόφαση που λάβαμε να συντάξουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. Κάποια σχόλια, σύντομα σχόλια, για κάποιες κατηγορίες σύνολα τροπολογιών. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω, λέγοντας καταρχήν ότι στόχος κάποιων από τις τροπολογίες είναι να έχουμε έναν πληρέστερο ορισμό της μικρής κλίμακας αλίας. Απαριθμώντας και κάποιες άλλες δραστηριότητες και κάποια άλλα τμήματα στόλου που και αυτά καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν στην έννοια της αλίας μικρής κλίμακας. Οι τροπολογίες αυτές συμπληρώνουν την αρχική εκδοχή της έκθεσης, την βελτιώνουν λοιπόν θα γίνουν λοιπόν αποδεκτές. Μια παρατήρηση όμως εδώ. Εδώ επαναλαμβάνουμε στις, κατά τη διάρκεια των 214 τροπολογιών έννοιες όπως η ερασιτεχνική αλία, η τοπική αλία, η παράκτια αλία. Νομίζω ότι καλό θα ήταν και αυτή ήταν και η πρόθεσή μας να το δούμε αυτό και με κάποιες από τις τροπολογίες που είχαν αρχικά ε, προταθεί για την έκθεση. Η έκθεση αφορά την ε, μικρή κλίμακα αλεία. Θα πρέπει λοιπόν από την αρχή να καθορίσουμε τι θεωρούμε ότι περιλαμβάνει η αλεία μικρή κλίμακα. Την αριστεχνική, την τοπική, κάποια ε, κομμάτια τη παράκτεια και μετά να αποφύγουμε την ποικιλία αυτή όρων ε, κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Να στην αναφέρουμε πάντοτε ως αλία μικρής κλίμακας, μικρή αλία. Έννοιες τις οποίες τα έχουμε αποσαφηνίσει από την αρχή, για να ξέρουμε τι συμπεριλαμβάνει ακριβώς αυτή η αλία μικρής κλίμακας. Είναι προτιμότερη αυτή η προσέγγιση από το να πολλαπλασιάζονται οι όροι κατά την ε, πρόοδο της έκθεσης, έραση τεχνική, ε, παράκτεια και ούτω καθεξής. Κάτι άλλο που θεωρώ επίση σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τι ιδιαίτερε ανάγκες της μικρής κλίμακας Αυτό επισημαίνεται και αρκετοί συνάδελφοι συμμερίζονται την αρχική μας παρατήρηση αυτή στην έκθεση. Βέβαια, κάποιοι ζητούν να απαλληθεί η μία αυτή. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να παραμείνει, διότι ήταν και σημείο αφετηρία για να ξεκινήσει η σύνταξη τη έκθεση αυτή. Θεωρούμε ότι η μικρή κλίμακα Ελία δεν καλύπτεται επαρκώ τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, που θα πρέπει να διατηρηθεί ιδίω στο σημερινό πλαίσιο τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική που δεν έχει ολοκληρωθεί. Και βεβαίω και ω ένα είδο προειδοποίηση για την ε, ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν επίση κάποια σημεία που δίνουν έμφαση στην, ε, στο ρόλο τη μικρή κλίμακα Αλίας βελτιώνουν και εξηγούν καλύτερα το τι αρχικά περιλάμβανε το πρώτο σχέδιο έκθεσης, νομίζω όλες αυτές οι τροπολογίες μπορούν να γίνουν ε, αποδεκτές. Σε ό,τι αφορά το σύστημα των μεταβιβάσιμων αδειών αλίας. Εδώ υπάρχει διαπίστωση, αναφέρεται η διαπίστωση, ότι ενέχονται κίνδυνοι με το σύστημα αυτό. Ναι, αλλά σε τι βαθμό οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ανατεχητιστούν, να αποφευθούν, να αντιμετωπιστούν. Αυτό είναι κάτι που διάφοροι συναδέλφοι το αντιμετωπίζουν με διαφορετικού τρόπου. Βεβαίω και ενέχονται κίνδυνοι, αυτό κανεί δεν μπορεί να το αρνηθεί. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τη διατύπωση που ε, προτείνουν μερικοί συνάδελφοι, ότι μπορεί να ενέχονται κίνδυνοι. Αυτό σίγουρα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τώρα το πώ θα αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι είναι κάτι άλλο που θα μα απασχολήσει σε άλλη φάση. Θα το σχολιάσω. Το θέμα τη ε, διαφοροποιημένη μεταχείριση με καθεστώτα και ε, συστήματα που να ε, προσαρμόζονται στι ανάγκε τη μικρή κλίμακα Εδώ υπάρχουν διαφορετικέ προτάσει, κάποιε αντιφατικέ μεταξύ του. Οπότε θα πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση, κάτι να επιλέξουμε Ίσως σε μια συνάντηση που θα οργανώ, ελπίζω να οργανώσω με τους σχεδόν εισηγητές. Ε, ίσως έτσι να καταλήξουμε σε μια συμμεπαστική πρόταση. Και για το θέμα αυτό. Ως προς τον ε, ορισμό της μικρής κλίμακας αλία, αλίας, εδώ πρέπει να ε, σκεφτούμε ποια επιλογή θα προκρίνουμε. Υπάρχουν διαφορετικές εντυπώσεις μεταξύ των οποίων θα μπορούσαν να επιλέγουν τα κράτη-μέλη. Κάποιοι λοιπόν προτείνουν την αρμοδιότητα για τον ορισμό την αναλάβουν τα κράτη-μέλη για να αποφασίσουν τι, τι συμπεριλαμβάνει και τι όχι η έννοια αυτή. Κάποιοι προειδοποιούν ότι καλό είναι να μην υπάρχουν ορισμοί που λαμβάνουν υπόψη είναι ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και σίγουρα κάποια επιλογή μεταξύ αυτών των διαφορετικών δρόμων θα πρέπει να γίνει. Έπειτα υπάρχουν Υπάρχει κάτι που άσχετα με το τι θέλουμε να συμπεριλάβουμε στον ορισμό και την απόφαση του αν θα ανατεθούν αυτά στα κράτη-μέλη ή όχι, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να λάβει και επιχειρησιακή διάσταση η έννοια αυτή. Τι σημαίνει δηλαδή ως προς την απόδοση δημοσιονομικών γραμμών από το Μελλοντικό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ε, συγκεκριμένες δηλαδή διατάξεις για την μικρή κλίμακα Αλία. Ε, απαριθμώνται κάποια κριτήρια, γίνονται συγκεκριμένε προτάσει που προτείνουν το να περάσουμε στα 15 μέτρα και άλλα κριτήρια όπως η διάρκεια των ε, αλληλευτικών ε, αποστολών. Κάποιοι προτείνουν τις 24 ώρες, κάποιοι περισσότερες ώρες, κάποιοι 12 μέτρα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω και να αποφασίσουμε και ω προ αυτά. Πάντω το σχόλιο ήθελα να το κάνω άσχετα με το ποια θα είναι η τελική μα επιλογή. Σε γενικέ γραμμές οι προτάσεις που γίνονται βελτιώνουν τα ισχύοντα κριτήρια της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή τέλο πάντων θα κάνουν λιγότερο αρνητικά. Ε, δεν είναι τόσο απλουστευτική, τόσο αρνητική προσέγγιση Όπω αυτή που μέχρι τώρα έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα είναι απαραίτητη λύση για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά αυτή η συζήτηση ελπίζω ότι θα γίνει για να εμβαθύνουμε στο όλο ζήτημα. Απλώ ε, το συγκρίνω με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το θέμα τη εγκύτητα. Κάτι που και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει στην έκθεση, ότι έχει να κάνει με την έννοια τη εγκύτητα, το πώ αυτή μπορεί να ενισχυθεί και επίση να δώσουμε έμφαση ότι αυτή καλύπτεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τι ιδιαίτερε ανάγκε τη μικρή κλίμακα αλεία. Εδώ υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που επιμένουν, επιβεβαιώνουν, ε, τονίζουν τη μεγάλη διαφορετικότητα των, του τι ισχύει στα κράτη-μέλη σε σχέση με την αλία αυτή, με αυτό το τμήμα στόλου. Οπότε αυτές οι τροπολογίες θα δείχνουν θετικής μεταχείρισης. Και όλα αυτά στο πνεύμα του να τονιστεί η διάσταση της εκείπητας και να μην έχουμε ένα σύστημα με ιδιαίτερα κεντρικό χαρακτήρα. Ως προς τις μεταβιβάσιμες άδειες αλλιώς. Δεν είναι εδώ αυτό καινούριο, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ακόμη και αντιφατικές. Δύσκολο να βρεθεί συμβαστική λύση, θα πρέπει όμως να επιλέξουμε τη μια ή την άλλη οδό. το να επιβληθεί υποχρεωτικά το σύστημα αυτό σε όλους είναι για κάποιους μια σκόπιμη λύση και για κάποιους άλλους όχι. Πάντως ο υποχρεωτικός χαρακτήρας, το να επιβληθεί αυτό, να είναι η μόνη διέξοδος, είναι κάτι που σε γενικές δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εγώ κατέγραψα ότι πολλές τροπολογίες μάλιστα τίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση ακριβώς. Όμως άλλες τροπολογίες αμφισβητούν αυτή την τοποθέτηση. Δηλαδή υπερασπίζονται το σύστημα αυτό, θέλουν να ισχύει υποχρεωτικά και να επιβληθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Eh, um, um, um- Μια προειδοποίηση εδώ. συμμερίζομαι την άποψη που εκφράζουν κάποιε από τι τροπολογίε ότι ορισμένε από τι παρατηρήσει που έχουμε κάνει εδώ για τη μικρή κλίμακα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα τμήματα. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να περιοριστούμε σε αυτό που τελικά, τελικά θα θεωρήσουμε ότι είναι η μικρή κλίμακα σαλία και να αποφύγουμε τις ε, πολυάριθμες αναφορές σε άλλα τμήματα στόλου. Αυτό μια μικρή διευκρίνηση ήτανε πέραν της ιδέας που πολλές φορές ε, υποκρύπτεται πίσω από κάποιες τροπολογίες ως προς το ζήτημα αυτό. Επίσης, κάποιες τροπολογίες ζητούν την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών ώστε να οριστούν τα τμήματα στόλου όπου υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα και να, να εντοπιστούν τα αίτια αυτής της πλεονάζουσας ικανότητας. Θεωρώ ότι πρέπει να στηριχθεί αυτή η ιδέα και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Θα γίνουν αποδεκτέ αυτέ τι τροπολογίε, κάτι που σημαίνει ότι βέβαια θα παληθούν άλλε τροπολογίε, όπω η 126 τη κυρία Φράγκα, που ζητούν την μείωση της πλευράς της του στόλου αναγκαστικά και μόνον βάσει των κριτηρίων της αγοράς. Βέβαια κάποιοι ζητούν το να εντοπιστεί πλενάζουσα ικανότητα ανατμήματα στόλου, κάτι που είναι εναλλακτική λύση όπως έλεγα προηγουμένως. Τώρα για τη στήριξη της ερασιτεχνικής αλίας. Να τονίσω εδώ ότι το πρόγραμμα στήριξης της ερασιτεχνικής αλίας δεν είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ούτε θα υποκαταστήσει τη λειτουργία του νέου ταμείου εδώ. Ούτε θετική διάκριση έχουμε εδώ βάσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη θάλασσα και την αλία, ούτε κάτι άλλο, απλώς θέλουμε μια καλύτερη διάρθρωση των εργαλείων που διατίθενται για τη θάλασσα και την αλία, προκειμένου να στηρίξουμε καλύτερα την μικρή κλίμακα αλίας και να διευκολυνθεί η χρήση από τα τμήματα αυτά του στόλου των διαφορετικών δυνατοτήτων που προσφέρονται. έστω και αν είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας Υπήρξαν λοιπόν προτάσεις να απαλληφθεί αυτό το πρόγραμμα στήριξης της μικρής κλίμακα αλίας. Εγώ νομίζω ότι καλό είναι να παραμείνει. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν, ούτε θέλουμε να υπάρχει ένα επιπλέον εργαλείο χρηματοδότηση πέραν των υπαρχόντων. Όχι, θέλουμε καλύτερη διάθεση, συνδυασμό και συνεργασία των υπαρχόντων εργαλείων, ώστε να προστατευτεί τελικά η μικρή κλίμακα αλία μέσα από τα ε, εργαλεία αυτά. Δράσεις χρηματοδότησης από το Μελλοντικό Ταμείο της Θάλασσας και Τη Αλία. Πολύ καλές προτάσεις. Πιστεύω ότι οι περισσότερες από αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ένα ζήτημα τίθεται σε σχέση με τον εξυγχρονισμό του στόλου. Προτείνεται να διαγραφεί η έννοια της ανανέωσης. Άλλοι προτείνουν να παραμείνει ο εξυγχρονισμός, άλλοι προτείνουν να διαγραφεί ο εξυγχρονισμός αλλά να παραμείνει η ανανέωση. θα πρέπει να επιλέξουμε. Εδώ τώρα για τις νομοδοτήσεις που μας έφτασαν από την Επιτροπή Επιφερειών και την ε, Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών θεωρώ ότι είναι νομοδοτήσεις ε, πλήρης που καλύπτουν το θέμα σε με ικανοποιητικό βαθμό. Απλώς μια προειδοποίηση. Θα μπορούσαμε να αποφελθούμε από ορισμένα σημεία και των δύο εκθέσεων για να τροφοδοτήσουμε την εκθέσή μας. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα σημεία και των δύο εκθέσεων, διότι έτσι θα χάσει την ισορροπία η δική μα έκθεση, διότι θα καταλήξουμε να μιλάμε τελικά από μια έκθεση για την μικρή κλίμακα κασαλία στη μικρή κλίμακα κασαλία για τι γυναίκε. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε δύο-τρει καθοριστικέ παραγράφου εδάφια από την κάθε έκθεση για να συμπληρώσουμε τα δικά μα λεγόμενα. Ήθελα λοιπόν να κάνω και αυτή τη διευκρίνηση ω προ Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πλήρε οι εκθέσει αυτέ και ενισχύουν ακριβώ το πνεύμα και τη δική μα έκθεση. Σημαίνω λοιπόν με ικανοποίηση την προσφορά του. Ευχαριστώ. Τέσσερι βουλευτέ ζήτησαν το λόγο. Πέντε, πέντε μάλλον. Ο κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χθε είχα ένα γεύμα εργασία. όπου παρευρέθηκε ο κύριος Φερέιρα, αντιπρόσωποι ΜΚΟ και της Κομισιόν. Πραγματικά βοήθησε και εμένα και άλλα μέλη της Επιτροπής αυτής να καταλήξουμε στις τροπολογίες αυτές και το, σημείο, το κεντρικό σημείο όλων των ε, συζητήσεων ήταν ο ορισμός της αλίας μικρής κλίμακας και είναι πραγματικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάτω από το ΕΤΘΑ και τις πιέσεις της Επιτροπής. Τα ωφέλη και, ε, της ε, νέας κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, είναι κυρίως στους στόλους μικρής κλίμακας. Ο τομέας αυτός απασχολεί περίπου 90.000 αλληλείς μικρής κλίμακας, ενώ ο τομέας μεγάλης κλίμακας απασχολεί περίπου 38.000 εργαζόμενους. Ο αριθμός λοιπόν των θέσεων εργασίας στα μικρά λιμάνια και στις ε, περιφερειακές τοπικές ε, κοινωνίες είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνο ε, ψαράδες, αλλά κάνουν και άλλες δουλειές. Είναι αγρότες, για παράδειγμα. Μέχρι τώρα, ο ορισμός της ελίας μικρής κλίμακας ήταν βασισμένος χονδρικά στο μέγεθος του σκάφους, περίπου 12 μέτρα ή κάτω από 12 μέτρα, χωρίς να χρησιμοποιεί ορισμένα εργαλεία, ε, χωρίς να είναι ε, μεταλλικά σκάφη ή από ατσάλι, συνήθως ξύλινα. Βέβαια τώρα χρησιμοποιείται και το fiberglass ως εργαλείο και τα σκάφη αυτά ε, ε, περνούσαν κάτω από 24, μέχρι μάλλον 24 ώρες στην θάλασσα. Αυτός ήταν ο ορισμός. Όμως εγώ πιστεύω ότι ο ορισμός αυτός πρέπει τώρα να συμπεριλάβει όλες τις έννοιες. Δεν πρέπει να είναι μόνο να περιοριστεί σε ορισμένα μόνο πράγματα. Ε, είναι πολύ αυστηρός ο ορισμός του σκάφος κάτω των 12 μέτρων. και αυτό να θεωρείται μικρής κλίμακας ελίας και να λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση από το ΕΤΑ. Θυμάμαι ότι ένας καπετάνιος μου έδειξε με μεγάλη περηφάνεια ε, πώς κόβοντας δύο μέτρα από το, ε, από το άκρο του πλοίου του, πώς το έκανα κατά από 12 μέτρα αυτή λοιπόν η προσέγγιση δεν μας βοηθά καθόλου, είναι σχεδόν γελία. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ορισμό ο οποίος να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που προενέφερα. Και νομίζω ε, μάλιστα ότι ο καιρός, ε, οι ώρες στη θάλασσα είναι ο πιο ε, ο ορισμός που μας βοηθά περισσότερο. Και πιστεύω πως αυτό που είδα για παράδειγμα στη Γαλλικία, όπου κάθε καπετάνιος έχει μια ειδική κάρτα και πριν βγει στη θάλασσα πρέπει να περάσει την κάρτα από μηχάνημα στην προκυμαία και η κάρτα αυτή με, το, με την πράξη αυτή αναγνωρίζει το σκάφος του, τον καπετάνιο, το πλήρωμα, τι θα κάνει, το είδος που θα ψαρέψει. Αυτό δίνει μια γενική εικόνα, αποτυπώνει το, το στιγμιότυπο αυτό στο, και το στέλνει στο αρμόδιο, στην αρμόδια υπηρεσία, στο αρμόδιο Υπουργείο. Επίσης όμως βοηθά, πιστεύω, και τον ορισμό της μικρής κλίμακας αλίας. Στην δική μου έκθεση προσπαθώ να προτείνω το, τη χρηματοδότηση του ΕΤΑ η χρηματοδότηση μάλλον αυτή να έχει βοηθητικό ρόλο και να υποβοηθείται και από την τεχνολογία. Χθε είχαμε εμπειρογνώμονε από την Ιρλανδία, οι οποίοι μα ενημέρωσαν για το πόσο ο οι μικροί στόλοι μπορούν να επηρεαστούν θετικά. Το ΕΤΑ, για παράδειγμα, πλήρωνε για ορισμένα εργαλεία στα μικρά σκάφη, τα οποία βοηθούσαν να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους και η κερδοφορία της ψαριάς τους. Η Κομισιόν μας είπε ότι το 75% της χρηματοδότησης θα προέρχεται από την Επιτροπή για στόλους μικρής κλίμακας με 25% συμβολή των κρατών μελών. Φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ ελκυστικό αυτό, αυτή η χρηματοδότηση και γι' αυτό είναι αναγκαίο ψηφίζοντας αυτές τις τροπολογίες να φροντίσουμε ο ορισμός να είναι ξεκάθαρος, έτσι ώστε να φροντίσουμε και για την χρηματοδότηση. Ευχαριστώ, κύριος Γκάλαχαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή για μια εκτενέστατη έκθεση φυσικά αποτελεί αυτό πλαίσιο για εμάς. Παρότι υπάρχουν σημεία στα οποία δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό και έχουμε και κάποιες τροπολογίες, έτσι κι αλλιώς. Μία από τις παραγράφους μου αρέσει ιδιαίτερα. Παράγραφος που αναφέρεται στη μικρή κλίμακα, στις μικρής κλίμακας αλληλεία και τη σύνδεσή της με τις παράκτιες περιοχές. Υπάρχει όλη η διασύνδεση με τον πολιτισμό, με την κουλτούρα των περιοχών αυτών και πάνω απ' όλα αναφέρεται στο γεγονό ότι αυτοί οι αλλοί επιστρέφουν κάθε μέρα στο σπίτι του. Δεν μπορούν να μείνουν στη θάλασσα πάνω από 24 ώρε. Στο τέλο τη βάρδια γυρίσουν. Αναφέρεται λοιπόν η διανυκτέρευση. Αν διανυκτέρευαν θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους αλλοί, ιδιαίτερα στον Ατλαντικό, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από την Βαλτική ή τη Μεσόγειο. Ο Ατλαντικός δεν είναι δεν έχει ασφαλείς θάλασσες σε σχέση με τις προηγούμενες. Μετά, υπάρχουν άλλοι παράγοντες για τα καύσιμα. Για παράδειγμα, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μετά, μιλάμε για, τις, ε, για την αλία μικρής κλίμακας. Δεν αναφέρεται τίποτα για τις απορρίψεις, για τα, τον τύπο των δικτυών που χρησιμοποιούν. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να το αναλογιστούμε ιδιαιτέρως για την, ε, όσον αφορά την στα πλαίσια της αναθεώρησης μάλλον της αλληλευτικής πολιτικής. Επίσης το ζήτημα των τοπικών αγορών. Δεν ε, προστίθεται κάποια οικονομική αξία αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θέλουν να αγοράσουν κατεψυγμένο ψάρι. Θέλουν, οι αγορέ προτιμούν το φρέσκο ψάρι και αυτό επίση πρέπει να αναφερθεί. Επίση, ένα πολύ σημαντικό θέμα ορισμό, στον ορισμό τη ε, της μικρή κλίμακα είναι πάρα πολύ απλό και θα διευκόλυνε την, ε, την διαχείριση για να, αν αναφερόμασταν μόνο στο μέγεθο, στα 12 μέτρα για παράδειγμα. Δεν είναι πλήρη όμω ο ορισμό αυτό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ας αντλήσουμε για παράδειγμα την ε, εμπειρία από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Είναι το μέγεθος ορισμό ορισμός σωστός. Όταν ψαρεύει κοντά στα, στην ακτή, ναι. Όταν ψαρεύεις όμως για παράδειγμα στι βορειοδυτικέ ακτές τη Ιρλανδία, όπου τα νερά είναι ταραγμένα, και ένα σκάφο μικρότερο των 12 μέτρων ε, μπορεί να καταστεί επικίνδυνο για το πλήρωμά του. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν μπορούμε επομένω μόνο να ορίσουμε την μικρή κλίμακα σαλία με το μέγεθο και να πούμε τελειώσαμε. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, ελπίζω όμως ο κύριος Φεραίρια να σκεφτεί αυτά που πρότεινα, και να τα θεωρήσει ρεαλιστικά, να εξετάσει τις τροπολογίες μου, ιδιαίτερα εκεί όπου αναφέρομαι στην Βορειοδυτική, Βόρεια Ιρλανδία, στη Βορειοδυτική Σκοτία και να αποφασίσουμε για έναν ορισμό της αλίας μικρής κλίμακας αφού έχουμε λάβει υπόψη τους καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα, στις επιμέρους ε, περιφέρειες της, ε, περιφέρειας αλίας. Επίσης, Οι περιοχές τις οποίες ανέφερα προηγουμένως που αντιμετωπίζουν άσχημε καιρικέ συνθήκες στον Ατλαντικό ε, αυτές δεν καθιστούν λογική την, λογικό τον ορισμό βάση του μεγέθους των 12 μέτρων. Επίσης, για τα μικρά νησιά που εξαρτώνται από την αλία, θα ήθελα να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν με κατανομή επιπλέον πόρων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτές οι μικρές κοινωνίες μπορούν να ευημερήσουν και να επιβιώσουν. Δεν μιλάω για μεγάλα μέρη, μιλάω για νησάκια 500-600 κατοίκων. Δεν έχουν άλλη επιλογή εκτός από την αλληλεία, αυτή τη μικρή αλληλεία. Πώς επιβιώσαμε στην Ιρλανδία το 1840 όταν έπεσε ο λοιμό. Με αυτά τα μικρά σκάφη καταφέραμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας. Δεν είχαμε άλλη απασχόληση. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να, να, να, να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτές οι κοινωνίες υπό τις παρούσες συνθήκες, εάν δεν, είχαν, εάν δεν έχουν την αλληλεία. Είναι μια πρακτική που στην Ιρλανδία ε, απαριθμεί εκατοντάδες χρόνια, αιώνες. Και όταν, εφόσον αναθεωρούμε την επιτυχία μας όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που έχουμε καταφέρει, πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτά τα μικρά νησάκια Επίσης, ε, για την πλεονάζουσα ικανότητα, δεν θα χάσω άλλο χρόνο. Θα προτιμούσα να, ακούσω, να, να δω τη λέξη έλεγχο. Και θα προτιμούσα να την ακούω τόσο συχνά όσο ακούω και την πλεονάζουσα ικανότητα. Αποφεύγουμε αυτό, αυτή τη λέξη, αυτόν τον έλεγχο. Μπορείς να έχεις ένα μεγάλο σκάφος. Εάν όμως συμπληρώσεις την ποσόστοσή σου για το μήνα ή για τη βδομάδα, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες αν συνεχίσεις να ψαρεύεις. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στον έλεγχο και την πλεονάζουσα ικανότητα. Επίσης, να πω στον κύριο Φερέρια ότι οι αλληλείς μικρής κλίμακας θα μπορούσαν να, θα μπορούσαν να του συσταθεί να γίνουν μέλη μεγαλύτερων ομάδων ε, συνεταιρισμός. Δεν είναι μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, δεν είναι μέλη ε, συνδέσμων παραγωγών και η βιωσιμότητα του κλάδου εξαρτάται από αυτό. Έτσι μπορούν να επιτύχουν ε, καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, για τα αλλιεύματα τους. Δεν είναι δική μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δική τους, όλων μας. Τους Αυτοί οι οργανισμοί τους αντιπροσωπεύουν και θα πρέπει να τους αντιπροσωπεύουν. Γενικά όμως πιστεύω ότι η έκθεση ήταν πάρα πολύ καλή και ε, φυσικά έχει περιθώρια βελτίωσης, αλλά ελπίζω να μπορέσουμε, βελτιώνοντάς την, να πείσουμε την Κομισιόν ότι να πείσουμε την Κομισιόν ότι πρέπει να λάβει υπόψη τους ε, αλληλείς μικρής κλίμακας. Κύριε Λόβιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή δεν είμαι η επίσημη σκιώδη συζητήτρια, ο συναδελφό μου Μπεσέινα. Μερικά σύντομα σχόλια όμως. Καταρχάς, όσον αφορά τον ορισμό της μικρής κλίμακας, συμφωνώ απόλυτα με όλους εσάς στο ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ χοντρικά φτιαγμένη. Τα 12 μέτρα δεν μας λένε κάτι. Έχει διαφορά. Πού είναι τα 12 μέτρα, στη Βαλτική, στον Ατλαντικό. Από την άλλη όμως δεν συμφωνώ και με ορισμένε προτάσεις τροπολογιών που προσπαθούν να καθορίσουν πιο συγκεκριμένα και περαιτέρω ε, ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, αλία ε, εντό 24 ωρών και αυτά τα ε, πρόσθετα κριτήρια. Προσωπικά πιστεύω ότι ο ορισμός της μικρής κλίμακας καλύτερο να γίνει ε, από το κάθε κράτος μέλος, γιατί διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία, με το είδος του αλλιεύματος, από κράτος σε κράτος, από τη... αλλιώς είναι στη Μεσόγειο και αλλιώς στη Βόρεια Θάλασσα. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά απλοποιημένο. Κάποια κράτη-μέλη πρότειναν τα 15 μέτρα αντί των 12 που είναι τώρα. Αυτό τα 12, είναι το 85% του ευρωπαϊκού στόλου τα 12 μέτρα. Αν πάμε στα 15, τι ποσοστό θα πιάσουμε, 95%? Θα υπάρχουν προτιμησιακές ε, συμπεριφορές εδώ και μεταχειρήσεις. Πιστεύω ότι τα πλοία, ανεξαρτήτως από το μέγεθός τους, μπορούν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Δεν είναι γνώμονας αυτό απόλυτος. Και αυτό επαναλαμβάνω κάθε φορά που συζητούμε αυτό το πράγμα για αυτή την έκθεση. Πολλές από τις προτάσεις σας με βρίσκουν σύμφωνοι. Αλλά για παράδειγμα, στη Σουηδία ήδη εφαρμόζονται κάποια πράγματα. Μπορούμε να το κάνουμε, να, να ε, δώσουμε προτιμησιακή πρόσβαση σε ορισμένα, σε τρία ναυτικά μίλια, σε δώδεκα ναυτικά μίλια. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ανακράτος κατά περίπτωση προσωρινές ελιευτικές δραστηριότητες είναι στο χέρι του κάθε κράτους μέλους να το ορίσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση, η κεντρική προσέγγιση, η συγκεντρωτική προσέγγιση. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν μ' αρέσει είναι η πρόταση ότι χρήματα θα πρέπει να δοθούν για, την, για τον εξυγχρονισμό του στόλου. Ο εξυγχρονισμό αυτός ο όρο τι εννοείται με αυτό, εννοείται την αυπήγηση νέων σκαφών και μου το επιβεβαίωσατε αυτό. Γιατί στη σουηδική μετάφραση υπήρξε μια σάφια. Η ναυπήγηση νέων σκαφών λοιπόν ε, είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα αντίθετη. Ακούσαμε την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου και είδαμε που οδήγησαν αυτές οι επιδοτήσεις και από τον Καντέκ και τον κύριο Καντέκ πριν, ο οποίος πρότεινε να υπάρξουν ε, πρημοδοτήσεις για τη διάλυση σκαφών. Θα μπορούσαμε και, να όμως τα χρησιμοποιήσουμε για να, να μικρότερα σκάφη. Υπάρχει λοιπόν, καθώς βλέπετε, κρυμμένη εκεί μέσα, επιχορήγηση για να ναυπήγηση νέων σκαφών και πιστεύω πραγματικά θα ήταν λυπηρό να υποστηρίζαμε αυτή την πρόταση τη πρότασή σας, διότι εγώ πιστεύω ότι αυτό μας έφερε στην πολύ άσχημη κατάσταση της ευρωπαϊκής αλίας που αντιμετωπίζουμε σήμερα, την πλεονάζουσα δυνατότητα. Και αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να ανακάμψουν τα εχθιαποθέματα. Διότι αυτός που έχει να κερδίσει περισσότερο από την ανάκαμψη είναι η αλίες μικρής κλίμακας. Γιατί αυτοί υπέφεραν περισσότερο από την εξάντληση των ηχθιαποθεμάτων κοντά στις ακτές. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, οι, οι αλληλείς μικρής κλίμακας θα μπορέσουν μόνοι τους να βγάλουν τα προς το ζήν, να διαχειριστούν τη δουλειά τους. Εάν ε, δεν γίνει αυτό, τότε όλες, ε, με μάλλον γίνει αυτό, όλες οι έρευνες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δείχνει ότι θα αυξηθούν τα εισοδήματα, ότι θα, μεγαλώ, θα αυξηθεί η απασχόληση. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Νίλσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να είμαι σύντομος. Όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιφερειών, όπου είμαι πλήρες τακτικό μέλος, και τόνισα ότι το θέμα της μικρής κλίμακας ηχθειοκαλλιέργειας είναι σημαντικό. Στα βόρεια της Σουηδίας και της Φινλανδίας είναι μια αναπτυσσόμενη δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας είναι μέρος της ε, παραγωγής της αλληλευτικής και θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο και για την ανάκτηση αποθεμάτων. Δημιουργεί, όπως είπα, θέσεις εργασίας και <coughs> στηρίζεται και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όταν ιδίω αυτές οι μικρές κλίμακας βιτεχνίες μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις περιβιωσιμότητας που είναι το ζητούμενο. Θα ήθελα λοιπόν να μην το αμελήσουμε και αυτό το τμήμα της, ε, όλης, του όλου κλάδου της μικρής κλίμακας αλλίας. Ευχαριστούμε κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Φερέρα, γιατί από κοινού με την Περιφερειακή Επιτροπή, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, τάχθηκε υπέρ ε, των τροπολογιών που υπέβαλα σε σχέση με την ε, εκτετική υδατοκαλλιέργεια, την αστρακοκαλλιέργεια και ούτω καθεξής. Μία τέτοια α, η είναι πολύ βιώσιμη, δίνει πολλές θέσει απασχόληση ε, όχι μόνο στη Γαλλική αλλά και στη Σουηδία και τη Φιλανδία. Αυτό που αναφέρατε κύριε Φερέιρα α, περιλαμβάνει την περίληψη συγκεκριμένων ατμάτων ελευτικών στόλων ή ε, ειδών, ειδών ή τύπων αλίας. Αυτό το θέμα με 35 ψήφους υπέρ, μία αποχή σχεδόν ομόφωνα πέρασε στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, και επισημάναμε την έλλειψη στατιστικών πληροφοριών και δικτών που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε πορίσματα, να στηριχτούμε σε πορίσματα επιστημονικά για να καταλήξουμε σε οικονομικά και κοινωνικά συμπεράσματα. Επίσης δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ορισμό της ε, μικρής κλίμακας αλίας. Καλό είναι να περιληφθούν ε, κάποια στοιχεία διαχείρισης, ε, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες οι τοπικές, οι γεωγραφικές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αλίας, κοινωνικά, βιολογικά, ε, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και το καθεξής. Πολλά από τα σημεία αυτά περιλαμβάνονται στις συμβαστικές λύσεις βέβαια, στις συμβαστικές τροπολογίες. Το ίδιο και για τη διαφοροποιημένη μεταχείριση της ε, βιοτεχνικής ελίας, ε, της υδατοκαλλιέργειας, οστρακοκαλλιέργειας ε, στη Γαλλία, προκειμένου να είναι βιώσιμη αυτή η υδατοκαλλιέργεια. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα ειδικά προγράμματα και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα ειδικά προγράμματα δεν συνιστούν δημιουργία νέων μηχανισμών, αλλά ανακατανομή των υπαρχόντων μέτρων. Και συμφωνώ και με τον κύριο Στίβενσον, θα θέλαμε να περιλάβουμε τα προϊόντα βιοτεχνικής αλίας που πληρούν τις προδιαγραφές της βιωσιμότητας της κοινής αλληλευτικής πολιτικής και λόγω βέλτιση των πρακτικών θα μπορούσαμε να τύχουν και μια ειδική πιστοποίηση, να έχουμε μια ευρωπαϊκή σφραγίδα, ένα ευρωπαϊκό σήμα για τα προϊόντα βιοτεχνικής α, μικρής κλίμακος και ε, βιώσιμης εκτε, ε, εκτατικής και όχι εντατικής το καλλιέργεια. Λοιπόν, αυτά ως προς, ε, τα, ως προς τα διάφορα κονδύλια, πώς θα πρέπει να κατανεμηθούν και να διευκρινίσουμε και τον ορισμό της μικρή ε, μικρής κλίμακος αλίας. Η κυρία Μπιλμπάου, τελευταία μιλήτρια. Όπως και εχθές θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη θέση μου, ξεκινώντας με την τροπολογία 6, στην οποία απευθύνω έκλειση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια διάγνωση της κατάστασης και της ε, αλληλευτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού Στόλου. Κάθε φορά που λαμβάνω το λόγο για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής επιμένω. Χρειαζόμαστε αυτό το check-up και της αλληλευτικής πολιτικής, αυτή τη διάγνωση για να γνωρίζουμε με σαφήνεια ποιοι είναι οι στόχοι μας, τι θέλουμε να υλοποιήσουμε και προς τα που οδεύουμε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 hemos estado tantos años engañándonos que al final tenemos que adoptar otro tipo de medidas para poner las soluciones de verdad. Hecha esta reflexión, hecha esta reflexión diría que ε, confiamos, creemos... Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια, ε, ένας ορισμός της ε, μικρής κλίμακος αλίας, δεν ξέρω, θα την πούμε βιοτεχνική, θα την πούμε αεραστεχνική μικρής κλίμακας και αυτό που θέλουμε να πούμε στις τροπολογίες μας είναι ότι δεν θα πρέπει να στηρίζονται στα, στις διαστάσεις μόνο στο πόσα μέτρα α, είναι ένα πλοίο. Γιατί υπάρχουν σκάφη ελευτικά που προστατε, σέβονται το περιβάλλον, πραγματοποιούν παραδοσιακή αλεία, δημιουργούν α, τοπικές θέσεις απασχόλησης, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και ε, προβαίνουν σε μια δίκη κατανομή των κερδών, χρησιμοποιούν αλληλευτικά εργαλεία που προστεύονται το περιβάλλον, άσχετο αν είναι 12-15 μέτρα το μήκος τους. Δεν θα πρέπει το μήκος των σκαφών να είναι τόσο <clears throat> καθοριστικός παράγοντας. Επίσης, αν ε, η πλειοψηφία των ομάδων θα ταχθούν υπέρ ε, τη λήψη αυτού του κριτηρίου του μήκους των σκαφών, θα πρέπει τουλάχιστον να εξαιρούνται όσες, ε, όσες, αλίες, όσες ε, βιοτεχνικές αλίες χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή ε, αλλιεύουν με παραδοσιακό τρόπο. Ούτε για το 24 ώρες συμφωνώ. Έχουμε πλοία που μένουν στη θάλασσα πάνω από 24 ώρες, αλλά επαναλαμβάνω χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία, αλλιευτικά εργαλεία που προστατεύουν το περιβάλλον, οικοσύστημα. Το ίδιο ισχύει και για την, τον αλίευση. Ούτε και εκεί το κριτήριο των 24 ωρών ισοδυναμεί με την προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε πληροφο... θέλουμε ενημέρωση, πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, ορισμός με βάση πιο ευρία κριτήρια. Ευχαριστώ, ξέχασα το πω στην αρχή, ευχαριστώ τον εισηγητή, αλλά θα πρέπει να ενισχύσει λίγο το ρόλο της περιφερειοποίησης. Να επιμείνουμε στην ανάγκη της περιφερειοποίησης και στη συμμετοχή του ελευτικού κλάδου στο έργο αυτό. Ενισχύοντας φυσικά και το ρόλο των συμβουλευτικών ε, συμβούλων. Διάλυση, εξυγχρονισμός, περιφερειοποίηση. Διαφωνώ με τη διαπίστωση του κυρίου Στίβεζον ότι εξυγχρονισμός σημαίνει κερδοφορία. Πρώτα συγκρότηση για να δούμε αν με τις αποφάσεις μας θα καταφέρουμε να καταστήσουμε επικερδή την αλληλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα του παροπλισμού της διάλυσης είναι μία πιθανότητα, μία δυνατότητα για να συγκροτήσουμε τον ελευτικό στόλο και να δούμε αν όντω ε, οι ενισχύσει για τη διάλυση εξυπηρετούν την ανασυγκρότηση. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε μια γενική επισκόπηση και μια σαφή αντίληψη. Το θέμα του εξυγχρονισμού επίσης. Ε, θα πρέπει ο εξυγχρονισμός να συμβάλλει στην βελτίωση των ε, εργασιακών συνθήκων των ναυτικών και των ψαράδων. Δεν συμφωνώ με την γνώμη του κυρίου Φεραίρα ό,τι αφορά την γνωμοδότηση τη Επιτροπή Γυναικών. Το θέμα τη ισότητα ε, έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Θα πρέπει τέτοιου είδου ευαισθησίε να τι εμπεριλαμβάνουμε σε όλε τι πολιτικέ μα. Γι' αυτό και κατέθεσα τροπολογίε όπου μιλάω για την ανάγκη και οι γυναίκε να συμπεριλαμβάνονται στις μεταρρυθμίσεις ε, και σε όλα τα ταμεία. Γιατί αυτές πλήττονται από τις ε, αρνητικές συνέπειες που ταλανίζουν τους ε, αλληλείς. Μην αμελούμε το ρόλο των γυναικών. Αρκούν τρεις προτασούλες για να συμπεριλάβουμε αυτή τη σημαντική ευαισθησία της ισότητας των δύο φύλων και στην πολιτική αυτή. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, ο κύριος Κούπερ, ευχαριστώ. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός. Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι και πολύ απαραίτητο η παρέμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λίγες μόνο παρατηρήσεις. Καταρχήν να συγχαρώ τον συντάκτη της ε, έκθεσης που θα είναι πολύ χρήσιμη στις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση και τις τρεις νομοθετικές προτάσεις που έχουμε επιτάπητος, γιατί όλες αυτές οι νομοθετικές προτάσεις ε, επηρεάζονται από το θέμα της αλλίας μικρής κλίμακας. Καταρχήν, το θέμα της διαφοροποιημένης μεταχείρισης. Πολλοί είπαν ότι όταν μιλούμε για μικρής κλίμακας αλλίας ή όταν μιλούμε καλύτερα για την κοινή αλληλευτική πολιτική, μιλούμε για πολιτική, αλληλευτική πολιτική για έναν στόλο που θα εξυπηρετεί κυρίως τη, το μικρής κλίμακα στόλο. Για τέτοια πολιτική μιλάμε. Όποιος και θα είναι ο ορισμός της μικρής ε, κλίμακας. Μεταξύ 70 και 90% των σκαφών είναι μικρής κλίμακας. Οπότε ουσιαστικά η κοινή λευτική πολιτική είναι πολιτική για την αλία μικρής κλίμακας. Οπότε η λογική του διαφοροποιημένου καθεστώτος δεν είναι προφανής. Γιατί ελάχιστο είναι το ποσοστό που δεν αφορά τη μικρή ε, μικρή κλίμακα αλληλεία. Δεν είμαστε υπέρ ενό διαφοροποιημένου καθεστώτος, είμαστε υπέρ κάποιων στοιχείων που θα είναι διαφοροποιημένα, αλλά όχι το συνολικό καθεστώ τη ΚΑΠ. Και αν θέλουμε μια βιώσιμη και παραγωγική κοινή ελευτική πολιτική, ο βασικός δικαιούχο ε, και αυτό που θα υποφεληθεί περισσότερο, από τέτοια παραγωγική πολιτική θα είναι ακριβώ η μικρή κλίμακο αλία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θέλουμε κάποια στοιχεία για το στόλο μικρή κλίμακα, γιατί όντω έχει ιδιαιτερότητε και μεριμνούμαστε να ληφθούν υπόψη στα διάφορα εργαλεία που προτείνουμε, στου διάφορου μηχανισμού που προτείνουμε. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα των μεταβιβάσιμων αλλιευτικών αδειών. επειδή δεν εξαιρέσαμε την αλληλεία μικρή κλίμακα από, από την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματο ακριβώ γι' αυτό ιδιαιτερότητε τη μικρή κλιμακοσαλίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, συμφωνώ. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο. Η πρόταση ε, για το ΕΤΘΑ είναι σε μεγάλο βαθμό πρόταση για τη, για μικρή κλιμακοσαλία. οι περισσότερες διατάξεις ε, του Ταμείου Θάλασσα και Αλίας αναφέρονται στα πλοία, όχι στους ε, εργαζόμενους. Γιατί επαναλαμβάνω, 80 με 90% των αλευτικών σκαφών ε, πραγματοποιούν μικρή κλίμακο αλεία. Υπάρχουν κάποια σημεία που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη μικρή κλίμακο αλεία. Μία καινοτομία είναι η πρόταση για τον ορισμό των εθνικών ποσών. Ένα από τα κριτήρια είναι το μέγεθος ε, των σκαφών. τα περισσότερα μικρά σκάφη έχει ένας ε, κράτος ε, ε, θα έχει περισσότερο πιο μεγάλο εθνικό ποσό. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τη σημασία της μικρής κλίμακος e και του μικρού κλίμακος στόλου. Τώρα, για το ποσοστό που δίνουμε με βάση το ΕΤΘΑ, υπάρχουν σημαντικές διαφορές Βέβαια, επειδή θα υπάρχει εθνική συγχρηματοδότηση, ίσως δεν φανεί αυτό σε εθνικό επίπεδο, πάντως ε, απαλλάσσουμε τις ε, εθνικές αρχές από την συγχρηματοδότηση υψηλά ποσοστά. Το θέμα της, ε, του βαθμού συγχρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό σημείο. Και υπάρχουν και κάποια ειδικά μέτρα που αφορούν τα μικρά σκάφη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά. Του αλείς με ολιγομελή πληρώματα. Για παράδειγμα, ενισχύουμε την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων που ισχύουν για μικρές επιχειρήσεις. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ικανές να φροντίζουν τον εαυτό τους. Μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό, αλλά το ΕΤΣΑ περιλαμβάνει κάποια μέτρα ειδικά για τα μικρά σκάφη και τη μικρή κλίμακος αλία και για την ανασυγκρότηση ε, ή την επαναχρησιμοποίηση ελευτικών σκαφών για άλλους στόχους, μόνο μικρής κλίμακος ε, αλής είναι επιλέξιμη για τις ενισχύσεις του ΕΤΘΑ. Και τώρα, ποιος είναι αυτός ο στόλος μικρής κλίμακος αλίας. Διαπιστώνω ότι Ο καθένα έχει τη δική του ιδέα για το ποιο θα πρέπει να εμπίπτει στον ορισμό αυτό της μικρής κλίμακος αλεία ή των μικρών σκαφών. Συνένεση δεν υπάρχει. Η μόνη συσπήρωση έγκυται στην απόρριψη του ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρήθηκε είτε ομός, είτε ακατάλληλος, είτε αστείος. Για να δούμε εσείς τι θα προτείνετε λοιπόν. Εγώ εξήγησα πάντως ότι είχαμε διαβούλευση για πολλά στοιχεία της ΚΑΠ και για τον ορισμό της μικρής κλίμακος. Και καταλήξαμε στον ορισμό αυτό ακριβώ εξαιτία τη διάσταση, τη μεγάλη διάσταση απόψεων που διαπιστώσαμε. Και λάβαμε την απόφαση για τον ορισμό που προτείνουμε μεν, αλλά είμαστε ανοιχτοί για οποιοδήποτε εναλλακτικό ορισμό εφόσον πληρούνται κάποια σημαντικά κριτήρια. Για παράδειγμα, να είναι απλός ο ορισμός, εύχριστος, να μπορεί να ελέγχεται. Αναφέρθηκε το θέμα των καρτών, ηλεκτρονικών καρτών. Να υπάρχει συμφωνία φυσικά, να είναι συνενετικός ορισμός, πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Και εκεί είναι και το δύσκολο. Γιατί κάθε ψαρά σχεδόν έχει τη δική του γνώμη για το τι εστί μικρή κλίμακο αλεία. Επίση, είναι σημαντικό όταν κατανέμονται κοινοτικά κονδύλια να υπάρχουν συνθήκε ίσου ανταγωνισμού, ισότιμου ανταγωνισμού. είναι πολύ αόριστο φλου ορισμό που διαστρεβλώνουν τις συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού, καλύτερα να μην τον εφαρμόσουμε. Και έγινε συζήτηση για το κατά πόσο το ΕΤΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, και κάποιες ενισχύσεις ανασυγκρότησης, ανανέωσης ή ναυπήγησης. Η κόκκινη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προτάσεις της ήταν αν με την ενίσχυση. Θα αυξήσουμε την ικανότητα ή θα διατηρήσουμε την πλεονάσια ικανότητα. Αν η απάντηση είναι καταφατική, δεν θέλουμε ενισχύσεις που να ενισχύουν την πλεονάζουσα ικανότητα που ήδη υπάρχει. Αν όμως η ενίσχυση αφιερώνεται σε επενδύσεις για το πλοίο που ενισχύουν την ελευτική του ικανότητα, τότε δεν την εγκρίνουμε. Αυτό ήταν, επαναλαμβάνω, η κόκκινη γραμμή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση. Καλώ και να ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταγράφω τι διάφορε παρατηρήσει και μόλι είναι δυνατόν, δεν έχει γίνει ακόμα, ε, βάσει του προγράμματο και των προγραμμάτων των Μακετών ΔΕ θα κοιτάξουμε να συναντηθούμε με τους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εξεύρουμε συμβιβαστικέ. Ε, ε, λύσεις. Τώρα τρει σημειώσει σε σχέση με τα σχόλια που μόλις έγιναν. Όταν μιλάμε για μικρά σκάφη και για μικρή κλίμακας αλεία, μιλάμε για το 80% του ευρωπαϊκού στόλου. όντω. Αλλά το είπα και επιμένω. Δεν μιλάμε αντιστοίχω και για το 80% των αλλιευμάτων. Οπότε, όταν ε, λέμε ως πρόσχημα, προσχηματικά μάλλον ότι με αυτό το 80% καλύπτουμε τα περισσότερα σκάφη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αλλιεύματα που καλύπτουν από αυτό το 80% των σκαφών είναι πολύ λιγότερα. Άρα έχουμε συνεννοηθεί εδώ ότι πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι τα αποθέματα τα οποία θέλουμε να καλύψουμε. 80% λοιπόν των σκαφών ναι, αλλά όχι 80% των ε, πόρων, των αλλιευμάτων. Αυτή λοιπόν είναι μια παρατήρηση που έπρεπε να γίνει γιατί αρκετές φορές το ακούμε αυτό σαν να μιλάμε για το σύνολο του ευρωπαϊκού στόλου. Αυτό να μην το ξεχνάμε λοιπόν. Ο ρόλος των κρατών μελών. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως. Ήδη σήμερα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα και το περιθώριο ελιγμών για να υλοποιήσουν μέτρα που προστατεύουν, καλύπτουν, ε, υπερασπίζονται τα ιδιαίτερα, τις ιδιαίτερες ανάγκες της μικρής κλίμακας αλία. Όντως, αλλά η έκθεση αυτή δεν έχει σκοπό να αντιταχθεί σε αυτήν την συνήθεια. Να συνεχίσει να γίνεται αυτά από τα κράτη-μέλη, αλλά και σε επίπεδο κοινή αλληλευτική πολιτική, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα. Η κυρία Λόβεν μα είπε ότι τα κράτη-μέλη μπορούμε να ορίσουν την προσωρινή πάυση των ελεκτικών δραστηριοτήτων, αν θέλουν, και εάν έχουν σκοπό να προστατεύσουν κάποια απόθυμα. Όντω. Αλλά αυτό που λέω, και αυτό είναι και ο σκοπό μια από τι τροπολογίε που έχουν αποκληθεί, θα έπρεπε να προβλέπεται δυνατότητα να στηριχθούν και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσα και Αλία αυτέ οι προσωρινέ διακοπέ ή αναστολή ελευτική δραστηριότητα. Είναι ένα από του σκοπούς που καλύπτουν κάποιες τοπολογίες και θα πρέπει να δώσουμε στα κάτι μέλη μια άλλη ευχέρεια να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το σημαντικότατο εργαλείο, αυτό το σημαντικό μέσο διαχείρισης των αλληλευτικών πόρων με έναν τρόπο βιώσιμο, δηλαδή την προσωρινή αναστολή αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Μην ξεχνάμε ότι κατά διάρκεια των περιόδων αυτών πάυσης θα πρέπει να μπορούν να επιβιώνουν οι εργαζόμενοι του χώρου. Σήμερα δεν προβλέπονται κονδύλια λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ελπίζω ότι στο μέλλον ε, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό είναι και ένα από του στόχου μια συγκεκριμένη τροπολογία. Τώρα για την ανανέωση των εξυγχρονισμών του στόλου. Δεν νομίζω ότι αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι το αν θα δοθούν επιδοτήσεις ε, για την ανανέωση του στόλου ή όχι. Βεβαίως πρέπει να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα. Βεβαίω πρέπει να δούμε τι γίνεται με την πλεονάζουσα ικανότητα και τι ελήφθηκε προσπάθειε, όμω δεν είναι αντιφατικέ αυτέ οι δύο προσεγγίσει. Ορισμένε προποθέσει θα μπορούσαν να δοθούν και βοήθειε για την ανανέωση σε περιπτώσει που δεν υπάρχει πρόβλημα την πλεονάζωση ικανότητα λόγω χάρη. Και αυτό συμβαίνει. Μπορεί λοιπόν να διαφέρει πάρα πολύ η επίδοση των στόλων μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν κάνει ιδιαίτερε προσπάθειε και τα τελευταία χρόνια έχουν καταλήξει σε μέσο όρο στόλου πολύ χαμηλή πολύ λιγότερο ισχυρή από ότι άλλα κράτη-μέλη που δεν έκαναν καμία προσπάθεια προσαρμογή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα αποκλειστικών, οριστικών απαγορεύσεων, οποιονδήποτε μέτρων στήριξη. Κάποια κράτη-μέλη έχουν στόλου διαφορετική ηλικία, υπάρχουν λοιπόν διαφορετικέ συνθήκε που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και ακριβώ πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο να προσαρμοστούν οι ικανότητε και στου πόρου. Συμφωνώ με διαφορετικέ προτάσει που ακούστηκαν για την εκτατική υδατολικαλλιέργεια, για το θέμα των γυναικών, Απλώς η παρατήρηση μου σήμαινε ότι το αν συμπεριλάβουμε όλα τα εδάφια της έκθεσης της ε, Επιτροπής Γυναικών στη δική μας την έκθεση μπορούσε να χαθεί η ισορροπία. Να μην το επαναλαμβάνω τώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να απομονώσουμε μια, δύο, τρει παραγράφου που να δίνουν την διάσταση του φίλου που και εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να διαφαίνεται μέσα από την έκθεση. Έγινε άλλωστε μια σύντομη μνήμα, ίσω να ήταν υπερβολικά σύντομη, το παραδέχομαι, στον ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών. Ε, και στη δική μα την έκθεση. Επίσης, όχι μόνο στην έκθεση της ε, επιτροπή των Γυναικών, αλλά και αυτή των περιφερειών ακούγεται αυτό. Αλλά να αποφύγουμε τις πολλές επαναλήψεις. Θα κάνουμε τη σχετική προσαρμογή. Σε συνεργασία με του και συγκεκριτέ ελπίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια και ολοκληρώσω αυτό το σημείο, μπορούμε να διακόψουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Θα επανέλθουμε στις 3 με το σημείο 21, καταρχήν την έκθεση Ριβελίνη. Ραντεβού στις 3. Πώς